Buongiorno a Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε. Ξέρετε ότι σήμερα το πρωί έχουμε τρία διαφορετικά πάνελ συζήτησης και γι' αυτό θα πρέπει να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ως συνήθως Έχετε συνάδελφοι στο φάκελό σας το πρόγραμμα, την ημερήσια διάταξη. Έγιναν κάποιες αλλαγές, έχουν ήδη ανακοινωθεί οι αλλαγές αυτές και έχουν ενημερωθεί οι συνάδελφοι. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, η ημερήσια διάταξη θεωρείται δεκτή. Περνάμε τώρα στο σημείο 2, ανακοινώσεις του, της Προέδρου. Όπως γνωρίζετε λοιπόν σήμερα το πρωί έχουμε και μία δημόσια ακροάση για το θέμα της εκ νέου ε, και βιομηχάνησης ε, του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο τέλος του πρωινού από τις 12.45 και μέχρι τις 14.15 και ε, θα έχουμε ένα γεύμα και μία παρουσίαση την οποία θα κάνει ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΡΝΑ. Το γεύμα αυτό λοιπόν και η παρουσίαση θα γίνουν στην ίδια αίθουσα. Τα μέλη είναι φυσικά προσκεκλημένα στη συνάντηση αυτή που θα έχουμε με το ΣΕΡΝΑ. Περνάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ουσιαστικά δηλαδή την δημόσια ακρόαση για την εκ νέου ε, εκβιομηχάνηση του Νότου της Ευρώπης. Θα ήθελα πριν από οτιδήποτε άλλο να καλωσορίσω όλους εσάς και τους προσκεκριμένους και για μένα είναι τιμή να κηρύξω την έναρξη των εργασιών αυτής της ακρόασης. Χαίρομαι που βλέπω αρκετούς συναδέλφους σήμερα εδώ που έχουν έλθει για να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω ε, ιδιαιτέρως τον τέος Υπουργό Βιομηχανίας της Πορτογαλίας και τέος Υπουργό Οικονομίας, τον καθηγητή Αουγκούστο Ματέους, ο οποίος θα κάνει την εναρκτήρια ομιλία. Να ευχαριστήσω και τους εισηγητές μας, ομιλητές από τον πανεπιστημιακό χώρο, από τον βιομηχανία και από την κοινωνία των πολιτών που θα μας μιλήσουν ε, για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη βαθύτερη οικονομική της κρίση και οι χώρες του Νότου υποφέρουν από τις αρνητικές επιπτώσεις όπως το κλείσιμο των μονάδων παραγωγής που έχει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Ε, πρέπει να επιστρέψει η Ευρώπη στην παραγωγή, πρέπει να αρχίσει πάλι να παράγει ιδιαίτερα ο, ο νότος της Ευρώπης. Σε τρία τμήματα λοιπόν η ακρόαση αυτή. Το πρώτο τμήμα θα μιλήσει για τα κλάστερ και την εξειδίκευση, την ευφυή εξειδίκευση και πόσο μπορεί να συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα μιας συγκεκριμένη γεωγραφικής περιοχής. Το δεύτερο τμήμα έχει σαν στόχο την δημιουργία εγγυήσεων για μια υφόρο ε, εκβιομηχάνηση και το τρίτο θέμα είναι το ακαθόδες θέμα της χρηματοδότησης. Εμείς ε, θα το ονομάσουμε αυτό οικονομικά μέσα και εταιρικέ σχέσεις. Κάθε τμήμα θα συνοδεύεται ή θα αποτελείται από δύο-τρεις ε, ομιλίες και στο τέλος θα υπάρξει δυνατότητα ερωτήσεων. Υπάρχει και η έκθεση για την εκ νέου εκπιομηχάνηση της Ευρώπης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της αηφορίας. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Beauty Coffer, ο οποίος είναι εισηγητής της πρωτοβουλίας, η οποία μόλις τώρα ξεκινά. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω να ευχαριστήσω και τους συντονιστές των διαφόρων πολιτικών ομάδων, όλος ιδιαιτέρως, που συμφώνησαν να διοργανωθεί αυτή η ακρόαση. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω όλους τους ε, υψηλού κύρους καλεσμένους μας. Μιλάμε για την εκ νέου βιομηχανοποίηση της ε, Νότιας Ευρώπης. Αυτό το θέμα, αυτός ο τίτλος ενδεχομένως κάποιοι να θεωρήσουν ότι είναι υπερβολικά έντονος. Μπορεί να παρανοηθεί ενδεχομένως και να θεωρηθεί ότι αγνοεί την βιομηχανική δύναμη που υπάρχει στις νότιες χώρες. Αλλά δεν είναι ασφαλώς αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αναζητούμε στρατηγικές για να ενισχύσουμε την βιομηχανία όλος ιδιαίτερος στο νότο της Ευρώπης. Και αυτό στο συγκείμενο της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του πρασμένου έτους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιλαμβάνει έναν πολύ προβλημένο αν θέλετε στόχο αυτόν της ανάκαμψης της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε ό,τι αφορά το μερίδιο του 20% ως στόχο για το έτος 2020 για τη μεταπητική βιομηχανία της Ευρώπης. Επίσης, να σας πω ότι συμφωνήσαμε ότι ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερος φιλόδοξος. Είναι σαφές όμως και πασιφανές ότι ο στόχος αυτός αποκλείεται να επιτευχθεί χωρίς στρατηγικές τόνωσης της ε, βιομηχανίας της Ευρώπης σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια στρατηγική εξόδου από την τρέχουσα κρίση, ιδιαίτερα για τα μέλη της Νότιας Ευρώπης, χωρίς να δοθεί μια νέα τόνωση στην βιομηχανία. Αυτό λοιπόν αποτελεί κοινή ανησυχία, μιας και είναι κοινή η μοίρα μας. Αυτό που ωστόσο με εντυπωσίασε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι δεν αφιερώθηκε ειδικό κεφάλαιο στον νότο της Ευρώπης. Και ένα από τα θέματα που με απασχόλησαν σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του σχεδίου έκθεσης ήταν κατά πόσον χρειάζονται ειδικέ στρατηγικές, ειδικά μέσα για την ενίσχυση των κρατών μελών του Νότου και μάλιστα με άμεσο τρόπο προκειμένου να υπάρξει βιομηχανική ανάκαμψη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρότεινα τη διοργάνωση της ακρόασης προκειμένου να συλλέξουμε ιδέες από τις χώρες του Νότου για τις χώρες του Νότου προκειμένου να μας διαφωτίσετε. Είμαι πεπισμένος ότι με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε μια προσέγγιση η οποία θα συνδυάσει ανταγωνιστικότητα αλλά και βιωσιμότητα. Αυτές οι δύο βασικές αρχές, ξέρετε, δεν ε, είναι αντιφατικές. Δεν χρειάζεται να είναι αντιφατικές. Ο συνδυασμός τους θα ενισχύσει την βιομηχανία και την οικονομία. Είμαι πεπισμένος. Και αυτό που ψάχνουμε είναι όχι μόνο αρχές που θα μας καθοδηγήσουν εν γέννη, αλλά και ιδέες, πρακτικές ιδέες σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες που ακούγονται και, ξέρετε, ε, ακούγονται, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το καθεξής. Αλλά εμείς θέλουμε συγκεκριμένες ιδέες που θα λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα τώρα και στο εγγύς μέλλον οι πρακτικές προσεγγίσεις είναι αυτές που μας λείπουν, αυτές που ελπίζουμε να ακούσουμε από όλους τους εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε να μας διαφωτίσετε και ευχαριστώ και σας Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μπουτικόφερ. Ξεκινάμε με το πρώτο μέρος και δίνουμε το λόγο στον καθηγητή κ. Γκούστο Ματέους. Παρακαλώ. Καλημέρα, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση και θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω το 15 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου για να σας δώσω μία εικόνα των απόψεων κάποιου που διδάσκει εδώ και πάνω 40 χρόνια βιομηχανική πολιτική, μακροοικονομική πολιτική και μακροοικονομικά και για δύο χρόνια ήμουν και υπουργό Οικονομίας της χώρας μου. Στην παρουσίασή μου συμπεριέλαβα πολλές πληροφορίες, ε, δεν θα μπορέσω να τις παρουσιάσω όλες σε 15 λεπτά, γιατί δεν είναι δυνατό, αλλά θα προσπαθήσω να σας δώσω μόνο τις ε, ουσιαστικές πληροφορίες. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο όλοι μιλάνε για επαναβιομηχάνηση, ανανέωση, αναγέννηση της βιομηχανίας. Γιατί, διότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Σήμερα ζούμε σε μια παγκόσμια οικονομία πολλαπλών ταχυτήτων, όχι μόνο δύο. Βλέπουμε πολλές μεταβολές ε, που οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αξία. Καθώς και στις διαφορετικές δυναμικές των διαφορών οικονομιών, ειδικότερα των ε, οικονομιών των νέων αναδυόμενων χωρών. Αναφέρθηκα στις 15 ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι για να επιστρέψουμε στο μέλλον. Απλά όπως γνωρίζετε τα νέα κρατημέλη έχουν ένα πρόσφατο παρελθόν ανάδυση στην Ευρώπη και διαφορετική ιστορία τα τελευταία χρόνια. Από το 2002 μέχρι το 2012 στις 15 χώρες της δεύτερης και τρίτης διεύρυνσης χάσαμε 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αλλά δημιουργήσαμε πάνω από 6.500 6,5 εκατομμύρια συγγνώμη, θέσεις εργασίας, ε, υπηρεσίες πληροφοριών επικοινωνιών και επιχειρησιακές υπηρεσίες. Κατά βάση κοιτώντα τα νούμερα της βιομηχανίας δεν απέχουν ιδιαίτερα από αυτό που θα έπρεπε να αναμένουμε μετά από μια οικονομική παγκόσμια ύφαση και δεδομένη στις νέες οικονομίες που βασίζεται σε γνώσεις και σε πληροφορική. Ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η οικονομική κρίση έχει μια τεράστια οικονομική διάσταση φυσικά αλλά είναι και μια κρίση ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειδικότερα στι χώρε του Νότου τη Ευρώπη. Και οι αρχικές 15 χώρες ε, αντιστάθηκαν καλύτερα και είχαν λιγότερη ανεργία σε σχέση με τις υπόλοιπε οικονομίε της Ευρώπης. Αυτό αιτιολογεί αυτή την ιδέα εστίαση τη επαναβιομηχάνηση στην Νότια Ευρώπη. Αλλά φυσικά οι καταστρεπτικές πτυχές της κρίσης δημιούργησαν στην Νότια Ευρώπη, ειδικότερα στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, και στην Ιρλανδία που δεν είναι βέβαια χώρα του Νότου ουσιαστικά η καταστροφή υπέστησαν οι λιγότερο ανταγωνιστικές εταιρείε ε, σε θέματα παραγωγικότητας ε, τα συνολικά νούμερα είναι σαφώς πολύ πιο ενδιαφέροντα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Τα νούμερα το λένε καθαρά. Η δική μου θέση είναι λίγο πιο επιθετική από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα επιτευχθεί το 20%. Αυτή η ιδέα, κατά την άποψή μου, του να έχουμε έναν αριθμό ώστε να υποστηρίξουμε ρητά και τεκμηριωμένα έναν στόχο βιομηχανικής πολιτικής, αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως και η στρατηγική της Λισαβόνας δεν λειτουργήσε όσον αφορά τους εθελοντικούς της στόχους. Αν κοιτάξει κανείς ε, τα νούμερα από το 2000 μέχρι το 2012 τα πάντα έπεσαν αρκετά γρήγορα και κάτι εντυπωσιακό είναι ότι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη η Γαλλία η οποία φυσικά είναι κατά κάποιο τρόπο ταυτόχρονα και νότια και κεντρική οικονομία για την οικοδόμηση της Ευρώπης σαφώς επηρεάστηκε περισσότερο από όλες. Με τώρα 10% λιγότερο στη τομέα της ε, βιομηχανικής παραγωγής. Κοιτώντας ε, την κατάσταση τώρα μετά την κρίση μπορούμε να συγκρίνουμε τη Γερμανία με τις άλλες χώρες και σαφώς η Γαλλία και η Ιταλία σε σύγκριση με την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία υπέφεραν πολύ σε αυτό το, υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κοιτώντας ε, τι μειώθηκε στο, σε απώλειες ε, στη βιομηχανική παραγωγή και τι αυξήθηκε τα κέρδη στους τομείς των πληροφοριών και των υπηρεσιών ε, του τριτογενούς τομέα σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που βλέπετε εδώ στα διαγράμματα θα δείτε ότι το συνολικό ισοζύγιο είναι θετικό με μία εξαίρεση την Πορτογαλία και μπορείτε να δείτε πολύ σαφώς ότι και στην Ιρλανδία όπως και στη Γαλλία το συνολικό ισοζύγιο δεν είναι θετικό. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην Ευρώπη δεν καταφέρνουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ε, αναδιάρθρωση εντό εισαγωγικών για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας, το ΑΕΠ μας και τις προσδοκίες όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Και έτσι αυξάνεται η ενεργεία. Και έτσι η ανάπτυξή μας παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Δεν αφορά μόνο τη βιομηχανική παραγωγή. Αφορά το σύνολο της οικονομίας παρατηρείται τεράστιος παγκόσμιος κατακαιρματισμός και αποδέσμευση των αλυσίδων αξίας και αυτό υπονομεύει το ρόλο των διαφόρων τομέων. Υπονομεύει και αυτή η διαδικασία κοινή θα έλεγα αξίας. Δεν είναι δηλαδή μια διαδικασία ενός μόνο επίπεδου. Δεν είναι μια διαδικασία ανοίγματο των αγορών με τον παραδοσιακό, με τον κλασικό τρόπο της μακροοικονομίας. Πηγαίνει πιο πέρα από αυτό, εξετάζει περισσότερο την προσέγγιση αυτή που αντιμετωπίζουν τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας. Τι κάνουμε, δηλαδή διανέμε όλο και περισσότερο όχι προϊόντα, όχι εταιρείε, όχι τομεί, αλλά δραστηριότητε σε ολόκληρο τον κόσμο και ορισμένε δραστηριότητε δημιουργούν υψηλή αξία Άλλες ε, όχι. Ή δεν ε, δημιουργούν επαρκή αξία. Ειδικότερα ε, όταν έχουμε να κάνουμε με δημοκρατίες με πολύ ψηλές απαιτήσει για το περιβάλλον, τις κοινωνικές, τα κοινωνικά δικαιώματα και όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει να εστιαζόμαστε τόσο πολύ σε συγκεκριμένους τομείς ή στη βιομηχανική παραγωγή. Κατά την άποψή μου χρειάζεται μια νέα ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που θα λύσει μέρος του προβλήματος. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βιομηχανική παραγωγή ως κάτι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Εγώ δεν βλέπω υποστήριξη σε όλες τις εθνικές και διεθνείς τάσεις ε, για επιστροφή στο παρελθόν της βιομηχανικής παραγωγής. Η ανακοίνωση της Κομισιόν δεν αφορά αυτό και η επαναβιομηχάνηση δεν αφορά μια επιστροφή στο παρελθόν. Δεν είναι επανάσταση, ούτε αναγέννηση. Είναι απλά μια προώθηση ενός νέου μέσου για περιφέρειες, για χώρες, για υπερεθνικές ενώσεις, ε, για μια γενικευμένη βελτίωση τη βιομηχανική παραγωγή βάσει γνώσεων, καλύτερων ικανοτήτων, δημιουργικότητα, καινοτομία, ώστε να προσαρμοστούμε στην παγκοσμιοποίηση και στι αναδυόμενε οικονομίε ω μια πραγματική ευκαιρία για την πρόοδο. Η επαναβιομηχάνηση αν έχει να κάνει με επιστροφή, θα πρέπει να μιλάμε για επιστροφή στο μέλλον, σε ένα πιο δυναμικό οικονομικά κόσμο, όπου η βιομηχανία θα αποκτήσει ένα νέο νόημα κινητοποίηση γνώση, επιστήμη, τεχνολογιών, δημιουργικότητα, μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών, ώστε να ικανοποιήσει τι όλο και πιο διαφοροποιημένες απαιτήσει ε, και τη ζήτηση παγκοσμίω με περιβαλλοντική ευθύνη και αηφορία. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με την ιδέα ότι για να βγούμε από αυτή την κρίση ανταγωνιστικότητας ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο δεσμό μεταξύ ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής συνοχής και αηφορίας στις οικονομίες και στις κοινωνίες μας. Η αξία όλο και περισσότερο εξαρτάται από τη γνώση και την οργάνωση που υποστηρίζουν τη βιομηχανική παραγωγή και όχι από την απλή διαδικασία του να ξεκινάμε από πρώτες ύλες για να καταλήξουμε σε τελικά προϊόντα. Έτσι ήταν η βιομηχανική παραγωγή στο παρελθόν, δεν θα είναι έτσι στο μέλλον. Αυτό θέτει πολλές απαιτήσει για τη βιομηχανική πολιτική, διότι μας οδηγεί να, στο να αλλάξουμε σχεδόν τα πάντα στη βιομηχανική πολιτική. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις παραδοσιακές κατακόρυφες πολιτικές και να εστιαστούμε σε όλα αυτά για τα οποία μιλήσατε εσείς, τα κλάστερ, τις οριζόντιες πολιτικές, συνδυασμένες δράσεις μεταξύ βιομηχανιών, πανεπιστημίων, τεχνολογικών ιδρυμάτων αλλά με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και τρόπο ανοιχτό Η βιομηχανική πολιτική πρέπει να εστιαστεί στο πώς εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία θέσεις εργασίας, πώς θα καταφέρουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και όχι το πού θα δημιουργηθεί ανάπτυξη. Δεν έχει σημασία το πού. Και φυσικά θα πρέπει επίσης να εγκαταλείψουμε τις γενικές προϋποθέσεις, γενικούς όρους, γενικόλογους όρους. Ε, αυτοί οι όροι είναι που οδήγησαν την Ευρώπη σε πολλά παράδοξα. Όταν εκ των υστέρων αξιολογούμε όλες μας τις δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής στα διαρθρωτικά ταμεία, παρατηρούμε παράδοξα. Βάζουμε πολλά λεφτά, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανεπαρκή για τα λεφτά που έχουμε επενδύσει. Και σκοπό είναι όχι να επενδύσουμε περισσότερα. σκοπό είναι να επενδύσουμε πιο αποτελεσματικά, με περισσότερε πιθανότητε να επιτύχουμε του σωστού στόχου, με το σωστό τρόπο. Όταν μιλάμε, για παράδειγμα, στα διορθωτικά ταμεία για έγκριση μια μεθόδου προγραμματισμού βασισμένη στα αποτελέσματα, αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ στα σοβαρά οι γενικές συνθήκες, γενική όροι δεν είναι καλό οδηγό, Ο καλό οδηγό είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς γνωρίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ορμή που έχουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε καλά και να εγκαταλείψουμε αυτά που κάνουμε λάθος. Κατά την απόψη μου λοιπόν πρέπει να ενοποιήσουμε τις βιομηχανικές πολιτικές με τις περιφερειακές πολιτικές. Γίνονται πολλές παρουσιάσεις για αυτό το θέμα. Αν κοιτάξετε ε, στη μεθοδολογία, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστούμε φυσικά στον πυρήνα της ε, μεθοδολογίας ε, που προτείνεται, αλλά να μην καταδικάζουμε μια περιφερειακή ή εθνική οικονομία στο να μην μπορεί να εξισορροπήσει το παράδοξο του μεταξύ τι κάνουμε στις, στα πανεπιστήμια, στις επιστήμες, στην τεχνολογία και του τι κάνουμε σε θέματα συνεργασίας εταιριών, ανάπτυξη νέων διαδικασιών, νέων λύσεων. Σκοπός είναι, κατά την απόψή μου, να έχουμε τρεις προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι κεντρική προσέγγιση περιφερειακών πανεπιστημιακών συστημάτων ε, και οι άλλες ε, είναι ότι έχουμε πολλές επιχειρήσεις στην Νότια Ευρώπη που μπορούν να υιοθετήσουν νέες διαδικασίες, νέα υλικά, νέα προϊόντα και χρειάζονται επιστήμες και τεχνολογίες που παράγονται σε ολόκληρο τον κόσμο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι στα, και στα πανεπιστήμια, στα κέντρα τα τεχνολογικά που βρίσκονται στις συγκεκριμένες χώρες, στις περιφερειές τους και πολλά από τα πανεπιστήμια μας, πολλά από τα ερευνητικά μας κέντρα, τα ακαδημαϊκά μας κέντρα έχουν γνώση που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τοπικές εταιρείες. Και αυτές οι προσεγγίσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν. Κατά την άποψή μου λοιπόν πρέπει να, να ανοιγόμαστε όλο και περισσότερο δημοκρατικά για να βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση, να προσαρμοστούμε στην παγκοσμιοποίηση και να έχουμε περισσότερη παγκοσμιοποίηση και όχι να προσπαθούμε να μείνουμε στο περιθώριο ενώ μεταβάλλονται οι οικονομίες μας και ο κόσμος και να αγνοήσουμε αυτή τη μεταβολή. Έχουμε ένα πρόβλημα στην Ευρώπη κατά την άποψή μου και πιστεύω μπορώ να το αναφέρω εδώ. Κοιτώντας τον κόσμο, οι δικέ μας οικονομικές πολιτικές στην Ευρώπη ε, είναι πιο φιλελεύθερες από τις οικονομικές πολιτικές των αναδυόμενων χωρών στην Ασία, στην Ιαπωνία και φυσικά αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε να αντιμετωπίσω όταν ήμουν Υπουργό Οικονομία και ερχόμουν εδώ στι Βρυξέλλε και έπρεπε να εξηγήσω στου συναδέλφου μου γιατί η θέση τη Ευρώπη έπρεπε να είναι μια καλή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των παραγωγών και των συμφερόντων των καταναλωτών. Σε θέματα κλωστή φαντουργία, χάλιβα, σκαφών πλοίων, την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη πρέπει πάντα να προσπαθούμε να εξισορροπούμε ό,τι κάνουμε για να δημιουργήσουμε σταθερές ε, ε, εταιρείε και θέσεις εργασίας και το τι κάνουμε για να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα πρότυπα διαβίωσης του πληθυσμού μας. Δυστυχώς η Ευρώπη στο παρελθόν ε, προωθούσε περισσότερο τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με τα συμφέροντα των παραγωγών και των όσων προσφέρουν θέσει απασχόληση και φυσικά και τη βιομηχανία. Και αυτό έχει να κάνει με τη δυσκολία που έχουμε να εξισορροπήσουμε τι διάφορε πολιτικέ, την εμπορική πολιτική, την πολιτική ανταγωνιστικότητα και τι βιομηχανικέ πολιτικέ. Θα πρέπει λοιπόν να εξισορροπήσουμε όλα αυτά εκ νέου γιατί το μέλλον της Ευρώπης βασίζεται σε μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τους στόχους μας για το κοινό μας νόμισμα. Η κρίση του ευρώ είναι επίσης μια κρίση σαφούς παραβίασης των όσων διδάσκουμε στα πανεπιστήμια για τις αρχές της οικονομικής πολιτικής. Έχουμε ένα χαλαρό περιβάλλον για την νομισματική πολιτική και ένα δύσκολο περιβάλλον για την δημοσιονομική πολιτική. Χρησιμοποιούμε δύο μέσα το επιτόκια και το συναλλαγματικές για να ε, επιτύχουμε τον ένα στόχο, να διατηρήσουμε τις τιμές, ε, τον πληθωρισμό όσο πιο κοντά στο 2% και μετά προσπαθούμε να τα επιτύχουμε όλα μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν είναι εφικτό, δεν έχει συνοχή και θα οδηγήσει την Ευρώπη σε μια πολύ δύσκολη θέση. Όπως βλέπουμε και διαπιστώνουμε ήδη. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την επαναβιομηχάνηση στην Νότια Ευρώπη ως έναν πολύ σημαντικό στόχο αλλά επίσης πρέπει να, δείξουμε, να αποδείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να μην είμαστε απλά μερκαντιλιστές και ότι υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσουμε να ανοίγουμε τις αγορές να έχουμε πολύ σαφείς ανταγωνιστικούς κανόνες στις αγορές αλλά όλα αυτά μπορούν να γίνονται στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης συνοχής, μιας μεγαλύτερης εξορρόψης των διαφορών αυτών συμφερόντων. Και αυτή η λίστα δημιουργήσει πρόσθετη αξία και περισσότερε θέσει εργασία στο μέλλον. Η επαναβιομηχάνηση φυσικά ε, εντείνει τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε καινοτομία ή διαφοροποίηση. Ζούμε σε εποχές όπου η δημιουργικότητα ο πολιτισμός, η τεχνολογία είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη δημιουργία αξίας. Είναι το ίδιο σημαντική με την καινοτομία. Η τεχνολογία είναι επίσης πολύ σημαντική. Αλλά το να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, ε, την κουλτούρα μας για να εξαπλωθούμε σε διεθνείς αγορές με πολλά διαφορετικά προϊόντα είναι πολύ σημαντικό. Η σπουδαιότητα της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού και ο ρόλος του τουρισμού στην Ευρώπη είναι σαφώς ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί. Χρειάζεται μια τέτοια προσέγγιση. Ο τουρισμός δεν, είναι μόνο, δεν έχει μόνο τεχνολογική πτυχή, μπορεί να δημιουργήσει αξία θέσεις εργασίας ε, στον τομέα της δημιουργικότητας του πολιτισμού. Θα προσπαθήσω να τελειώσω τώρα όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό που ήθελα να πω. Εγώ θα ξέχναγα το 20% όσον αφορά τη συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ. Διότι κάτι τέτοιο μπορεί να μας οδηγήσει σε υψηλότερη συμβολή στο ΑΕΠ από τη βιομηχανία, αλλά μειωμένο ΑΕΠ στην Ευρώπη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νέα συνεργασία στη βιομηχανική παραγωγή για να δημιουργηθεί ΑΕΠ νέο Σήμερα έχουμε πολλές βιομηχανίες και υπηρεσίες. Έχουμε πολλές υπηρεσίες εντός των βιομηχανιών και πολλή βιομηχανία στις υπηρεσίες. Αν δείτε την οικονομία που βασίζεται σε γνώση, ανθεί στις, παραγωγή, στις πρωτεύουσες παραγωγές. Αν δείτε πολλά πρωτεύοντα προϊόντα βλέπετε ότι, χάνετε, ότι χρειάζεται γνώση. Σήμερα πια δεν φτιάχνουμε κρασί στην Ευρώπη απλά μετατρέποντας τα φιλιά σε μουστο το κρασί παράγεται μετά από μελέτη της γεύσης, της αηφορίας και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι γνώσεις και τα πανεπιστήμια. Οι γνώσεις αυτές χρειάζονται για να δημιουργήσουν αξία με έναν νέο τρόπο. Η σπουδαιότητα της βιομηχανικής παραγωγής είναι ότι δεν μπορεί να αποφύγει κανείς να κάνει πράγματα μέσω της βιομηχανίας. Έτσι ήταν πάντα και έτσι θα είναι πάντα. Ο τρόπος αποτελεσματικός παραδοσιακός τρόπος χρήσης των υλικών, επεξεργασίας των μετάλλων, νέοι τρόποι εξευγενισμού του, του πετρελαίου, εξευγενισμού των ελαίων. Αυτό είναι ο ρόλος της βιομηχανίας, αλλά η βιομηχανία όλο και περισσότερο θα βασίζεται σε γνώσεις, στις ικανότητες εφαρμογής νέων αποτελεσματικών διαδικασιών και νέων προϊόντων. Αυτό μας αναθέτει κάποια καθήκοντα τα οποία θα μας οδηγήσουν να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες μας ε, στην Ευρώπη. Ε, καθήκοντα, εργασίες που θα προσθέσουν αξία με συνεργατικό τρόπο, με συνεργασία μεταξύ πολλών διαφορετικών θεσμών και οργανισμών. Τα μέλη αναφέρουν ε, ρητά τα προβλήματα στην Νότια Ευρώπη η ανταγωνιστικότητα πληρώνεται με ισχυρό τμήμα στην, τίμημα στην Νότια Ευρώπη και όπως είπα σαφώς σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία όπως και σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου η διαδικασία προσαρμογής ε, ήταν εξαιρετικά δύσκολη και δύσκολη στη διαχείριση όχι μόνο φυσικά από τους Έλληνες μόνο αλλά κοιτώντα αυτή τη Γερμανία που λάμπει στην Ευρώπη και συγκρίνει κανείς τη Γερμανία με άλλες χώρες στον κόσμο θα δει ότι ακόμη και η Γερμανία δεν λάμπει τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στον κόσμο τα πράγματα κινούνται εξαιρετικά γρήγορα. Συνεπώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Νότιας Ευρώπης αλλά και ολόκληρη της Ευρώπης. Και έτσι χρειαζόμαστε πολλές διαφορετικές λύσεις. Κάτι που πρακτικά που ξέχασα να πω σε πρακτικά θέματα είναι ότι χρειαζόμαστε λειτουργία της αγοράς σε θέματα αξίας και όχι σε θέματα νούμερων και προϊόντων. Η αξία μιας εταιρείας είναι το τι πουλάει μια εταιρεία. Και αν και δούμε τη Γερμανία, όπου οι καλύτεροι επιδόσεις ε, όπου παρατηρούνται καλύτερες επιδόσεις μείωση των τιμών και αύξηση των εξαγωγών Ε, στις νότιες οικονομίες όπως στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία τα πράγματα δεν ήταν πολύ διαφορετικά από τη Γερμανία και στη Σουηδία την οποία δεν την περιέλαβα διότι δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης βλέπετε εδώ πολλές πληροφορίες απλά ήθελα να σας υπενθυμίσω κάτι τι είναι σημαντικό στις παγκόσμιες εξαγωγές ότι Εδώ ουσιαστικά βλέπετε διαφορές εξειδίκευσης ε, και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ε, οι ακαθαρίστες εξαγωγές και η προσθέμενη αξία είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ σε ακαθαρίστες εξαγωγές έχουμε εισαγωγές ε, και εξοπλισμό των πόρων και εθνική προστιθέμενη αξία. Η Ευρώπη πρέπει να εξεταστεί το πράγμα υπερεθνικά και το πώς θα συμμετέχει στην παγκοσμιοποίηση για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της. Και οι προσδοκίες της είναι η προστιθέμενη αξία. Και εδώ όσον αφορά την προστιθέμενη αξία βλέπετε εδώ το περιεχόμενο των εισαγωγών σε διάφορες ευρωπαϊκές οικονομίες. Όπως βλέπετε έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλά σε αυτό το τομέα. Μπορεί κανείς να βελτιώσει τις σχέσεις του οικοδομώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχετε στο νου σας μια προτίμηση προς την Ευρώπη, όχι νομική προτίμηση, αλλά να συνεργαστείτε ώστε να δημιουργήσετε αξία στην Ευρώπη. Και πολλά μπορούν να γίνουν όχι σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία των εξαγωγών μας. Και θα ολοκληρώσω με τρεις ε, προτάσεις, συστάσεις. Πρακτικά θα πρέπει να λύσουμε τη διαρθρωτική μας κρίση ανταγωνιστικότητας με τρεις τρόπους. Βελτίωση της ε, παραγωγής προϊόντων αξίας. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι οι νότιες οικονομίες ε, δεν είναι ότι έχουν το πρόβλημα της αποτελεσματικότητας, αλλά ότι οι θέσεις τους αυτών των οικονομιών είναι κατακαιρματισμένες όσον αφορά τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και προμηθειών. Πρέπει να γίνει δηλαδή να δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση της ποιότητας και όχι της ποσότητας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων, όπου μπορούμε να είμαστε πολύ επιλεκτικοί. Δεν είναι το πρόβλημα η παραγωγικότητα. Το πρόβλημα είναι πολλά, ο συνδυασμός πολλών πραγμάτων και η συνεργατική προσέγγιση είναι εύκολο λοιπόν, αν θέλει κανείς πρακτικά να φέρει αποτελέσματα, πολύ επιλεκτική επιλογή των κονδυλίων και συνεργατική εφαρμογή. Ας κάνουμε με τις εταιρείες ό,τι κάνουν και τα πανεπιστήμια μεταξύ τους. Ας συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε πραγματική αξία. Η ανάπτυξη λοιπόν και συντελεστών ε, ανταγωνιστικότητας ε, είναι κάτι σημαντικό για την Ευρώπη. Πρέπει να πουλήσουμε στον κόσμο και στους πληθυσμούς μας ε, μέσω των οικονομικών μας δραστηριοτήτων αυτά που έχουμε δημιουργήσει και όχι αυτά που έχουμε αγοράσει. Πρέπει να πουλάμε τις δικές μας γνώσεις, τη δική μας δημιουργικότητα, τη δική μας ποιότητα, τη δική μας ικανότητα να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα και νέες λύσεις για την αγορά. Τέλος, Χρειαζόμαστε μια πιο εντατική, πιο ευφυή, χρησιμοποιείται πολύ σήμερα αυτός ο όρος ευφυής, πρέπει να είμαστε πιο ευφυείς όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι κίνητρο, δεν είναι ούτε η αιτία των προβλημάτων μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ηγηθούμε αυτής της παγκοσμιοποίησης γιατί αυτή είναι η ιστορία της Ευρώπης τώρα δημιουργεί έναν μεγάλο παγκόσμιο κόσμο και όχι ένα μικρό κόσμο Ας μην ξεχνάμε μικρές χώρες του Νότου όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία που κάποτε χώρισαν τον κόσμο στα δύο. Μη φοβόμαστε λοιπόν την παγκοσμιοποίηση. Αλλά χρειαζόμαστε τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν στην παγκοσμιοποίηση με το ισχυρό της νόμισμα η Ευρώπη για παράδειγμα δεν ε, επένδυσε ιδιαίτερα στον κόσμο. Μια, οικονομία, μια ομάδα οικονομιών που δημιουργούν ένα ισχυρό διεθνές νόμισμα και δεν επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στον υπόλοιπο κόσμο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αποτελεί μυστήριο. Ένα ισχυρό νόμισμα χρησιμεύει μόνο αν το επενδύσει κανείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Ματέους για την παρουσίασή του, αν και χρησιμοποίησε δύο φορές το χρόνο τον οποίο είχε στη διάθεσή του. Θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Καρβάλιο προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή κύριο Ματέους η παρουσίασή σας ήταν ενδιαφέρουσα και σημαντική. Να μας μιλήσετε λίγο για τη σχέση ανάμεσα στην επένδυση στην γνώση και στην οικονομική ανάπτυξη. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν αρκεί κανείς να επενδύει στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Εμείς στην Πορτογαλία έχουμε επενδύσει στην έρευνα, έχουμε επενδύσει στην εκπαίδευση, αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην οικονομία. Και αυτό ίσως να ισχύει και για πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Απαιτούνται πολύ περισσότερες προϋποθέσεις, κάποιες από αυτές αναφερθήκατε, μακροοικονομικές λειτουργία της αγοράς κτλ και τότε μόνο η ε, γνώση αντικατοπτρίζεται στην οικονομία. Αν όμως οι προϋποθέσεις ε, είναι καλές. Τι είναι αυτό το οποίο θα καταστήσει τις γνώσεις μας εδώ στην Ευρώπη ε, και θα τις κάνει προϊόντα και προϊόντα τα οποία η Ευρώπη θα εξάγει. Ξέρετε ότι τα φωτοβολταϊκά σαν παράδειγμα εμείς τα αναπτύξαμε, άλλοι τα παράγουν ποιος είναι ο παράγων αποτελεσματικότητας που μας λείπει έτσι ώστε η μεταποιητική αυτή η κατασκευαστική βιομηχανία να μείνει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα και αυτό θα δημιουργήσει απασχόληση. Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι η είναι η ύπαρξη ενός εξαιρετικού πανεπιστήμιου. Η Ντέμπλερ είναι στη Στουτγάρδη επειδή στη Στουτγάρδη υπάρχει και ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Εκεί όπου υπάρχουν εξαιρετικά πανεπιστήμια υπάρχουν και ιδιαίτερα έντονες οικονομικές ζώνες παραγωγής. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Σύντομα. θα πρέπει να είμαστε επακριβέστεροι ε, για τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στην έρευνα και την καινοτομία. Προφανώς η έρευνα στρέφεται στην επιστήμη, κοιτάει την επιστήμη, η καινοτομία κοιτάει την αγορά. Η έρευνα είναι απλή, η καινοτομία είναι περίπλοκη. Πάρα πολύ συχνά στην Ευρώπη και στις νότιες χώρες ασχολούμεθα με την καινοτομία αλλά κατά κάποιο τρόπο έχουμε, προκαταλαμβάνουμε τις ανάγκες της αγοράς. Το θέμα είναι να ασχοληθούμε με την καινοτομία έχοντας όμως υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής θα μάθουμε πολλά ιδιαίτερα από τις Ηνωμένε Πολιτείε που χρησιμοποιεί το δημόσιο χρήμα για τη διάδοση της έρευνας της πληροφορίας, της ενημέρωσης, έτσι ώστε το περιβάλλον των μικρομεσαίων να εμπλουτίζεται και να λειτουργεί καλύτερα. Δεύτερον, πράγματι η επιστήμη είναι ένα καθολικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι το περιφερικό. Το περιεχόμενα της επιστήμης είναι σφαιρικού παγκόσμιου χαρακτήρα. Ενώ η χρήση σε καθημερινή βάση γίνεται τοπικά η παγκοσμιοποίηση μπορεί να ενισχύσει την εδαφική τοπική ανάπτυξη για τη δημιουργία πλούτου και θέσεων απασχόλησης. Όμως τα τοπικά πανεπιστήμια, ακόμα και τα πολύ καλά πανεπιστήμια, πρέπει να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην παγκόσμια γνώση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν περιοριστικές περιφερικές μορφές περιορισμού. Εάν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς στην Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργήσουμε ορισμένες περιφέρειες τις οποίες τα πανεπιστήμια θα είναι εξαιρετικά και θα συνεργάζονται με εξαιρετικές επιχειρήσεις όχι για τους εαυτούς τους αλλά για τους πολίτες. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ακριβέστεροι σε σχέση με τις ανάγκες της οικονομικής πολιτικής και της βιομηχανικής πολιτικής. Το, θέμα, το θέμα δεν είναι να διαφημιστούμε στους δημοσιογράφους και στα μέσα ενημέρωσης. Το θέμα δεν είναι να λαμβάνουμε πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις μόνο για τις ειδήσει των οκτώ. Θα πρέπει να προωθούμε θέσεις και να δημιουργούμε μέσα σε 24 ώρη βάση και με πραγματική προστιθέμενη αξία. Έτσι με πραγματικές επιχειρήσεις, με πραγματικούς ανθρώπους θα παράγουμε την αξία που απαιτείται σε παγκόσμιο επίπεδο όπως ζητούν οι καιροί και θα βελτιώσουμε και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα που παράγουν την γνώση, γνώση όπως είπα που θα ενσωματώνεται από τους πολίτες, θα κερδίζουν όλοι από αυτήν και έτσι θα διαμορφώνονται οι οικονομικές πολιτικές με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βοηθούνται οι επιχειρήσεις σε επίπεδο γνώσεων, σε επίπεδο εμπειρεών όχι μόνο εξοπλισμών το θέμα δεν είναι να αγοράζει κανείς νέα μηχανήματα και να πατάει το κουμπί και από την άλλη να χάνει τη φαιά ουσία της γυραιάς υπήρου προς άλλες χώρες και περιοχές. Είναι θέμα πολιτικής ευθύνης και είναι και θέμα πολιτικού θάρρους. Ευχαριστώ τον καθηγητή Ματέους για την διευκρίνηση αυτή. Θα μιλήσουμε τώρα για τα κλάστερς και τους πόλους ανταγωνιστικότητα. Ο κύριος Μακιός έχει το λόγο για 10 λεπτά. Να σας ζητήσω παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να περάσω κατευθείαν σε μία απτή λύση για το πρόβλημα το οποίο ανέφερε η κυρία Καρβάλιο. Τα κλάστερς οι συνεργατικοί σχηματισμοί αποτελούν ένα εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη και κοιτώντα τα θέματα τη καινοτομία. Η καινοτομία σήμερα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Επειδή αποτελεί μια ευφυή ιδέα, η οποία όμως θα μετατραπεί σε προϊόν. Αυτό είναι ο σκοπός και το εργαλείο για να το αποτύχουμε αυτό είναι τα clusters. Και σκεφτείτε την προσέγγιση της Silicon Valley που άλλαξε τον ε, κόσμο. Σκεφτείτε το Skype σε ό,τι αφορά την Εσθονία, την Φιλανδία, τα συστήματα τα καινοτομικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση που κατέστη ηγετική σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα τεχνολογίας. Τι κάνουμε λοιπόν στην ε, πρωτοβουλία Coralia Clusters στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια ήταν καταλητικός ο ρόλος μας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομία και της περιφερειακής ανάπτυξης. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Δίνουμε στους νέους τη συμμετοχή στην ανάπτυξη της χώρας και ένα όραμα ασφαλώς, ένα όραμα στην Ελλάδα και αλλού ασφαλώς. Στην ε, Μεσόγειο πριν από 2.500 χρόνια οι Έλληνες άλλαξαν τον κόσμο, τη μορφή του κόσμου χάρη στην έννοια της αγοράς. Ένα κλάστερ, ε, μια, ε, ένας χώρος ομαδοποίησης όπου ο κόσμος συνερχόταν για να συζητήσει την ιονική φιλοσοφία. Ο Περικλής, ο Ευκλήδης, τη γεωμετρία, ο Αρχιμίδης, ε, τη μηχανική ο Πλάτων την ανθρώπινη συμπεριφορά, ο Αριστοτέλης, χρησιμοποίησε τον κόσμο της ελληνικής γλώσσας και άλλαξε τη μορφή του κόσμου με την πρώτη, αν θέλετε, παγκοσμιοποίηση. Δίνουμε λοιπόν ένα όραμα στο νέο. Ένα στόχο, το στόχο της κοινοτομίας, της σχεδίου, του σχεδιασμού στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία ή οπουδήποτε αλλού. Και γιατί? Γιατί σήμερα με το διαδίκτυο μπορούμε περιφερειακά να αναπτυχθούμε και να α, είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι είναι λοιπόν τα κλάστερς ε, αναφέρθηκε στο παρελθόν ότι πρόκειται για γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεμένων ε, ανεξαρτήτων ε, εταιριών και θεσμικών οργάνων, πανεπιστημίων δηλαδή, σε ένα συγκεκριμένο τομέα ένας πυρήνας, δηλαδή μια οικονομία κλίμακας λοιπόν, συνεργασία μεν, αλλά και συμπληρωματικότητα. Αυτές είναι οι βασικές λέξεις, οι λέξεις κλειδιά. Και θεωρώ ότι στην δημιουργικότητα έγινε και η χαρά της δημιουργίας. Αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει να επανέλθουμε στην δημιουργικότητα ως πηγή απόλαυσης, χαράς. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να εξέλθουμε από τη δύσκολη κατάσταση. Η βιομηχανία, η έρευνα, η ανάπτυξη, όλα αυτά θα πρέπει να συνεργάζονται. Τι κάνουμε λοιπόν στο πρόγραμμα Κοραλία. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημά μας. Πρόκειται για ένας καταλήτης που συνενώνει τον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά και τους δημόσιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους χρηματοδότης, τις τράπεζες, δυστυχώς αλλά και τα επιχειρηματικά κεφάλαια, αλλά και ασφαλώς ε, τα μέσα ε, αγοραστών, ε, τις δομές υποδομής. Γίνεται καταρχάς μια καταγραφή του τομέα μια προπαρασκευαστική εργασία. Λέμε ότι έχουμε 10 ε, εταιρείε οι οποίε, για παράδειγμα, μπορούν να δραματίσουν ένα ρόλο στην μικροελεκτρονική. Με αυτή τη χαρτογράφηση περνάμε στην πρώτη φάση. Εφαρμογή δηλαδή και εξέταση κατά πόσον μπορούν να συνεργαστούν αυτέ οι εταιρείε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κατά πόσον μπορούν να συνεργαστούν και να παράγουν από κοινού. Και μετά φέρνουμε σε επαφή τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια. Χρειαζόμαστε ασφαλώ και χρηματοδότηση για να αποδεχτεί κατά πόσον αυτό το σύστημα, το οικοσύστημα μπορεί να συνεργαστεί, να παράγει αγαθά που θα παράγουν τελικά πλούτο για την Ευρώπη και για τη χώρα. Σε έξι χρόνια λοιπόν το πρόγραμμα Κοραλία δημιούργησε ένα μικρό θαύμα για την Ευρώπη. Δημιουργήσαμε ένα κλάστερ μικροηλεκτρονικής που σήμερα περιλαμβάνει 130 μέλη, 80 εταιρείες 40 πανεπιστημιακά ιδρύματα και περιφερειακά ιδρύματα, όπως το EPR, δικηγόρους και το καθεξής. Και εδώ και δύο χρόνια έχουμε και ένα νέο κλάστερ στην ε, τεχνολογία του διαστήματος και άλλο ένα κλάστερ, άλλο ένα συνεργατικό σχηματισμό σε ό,τι αφορά το gaming, ε, τα τεχνολογίες avatar και το καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το οικοσύστημα τριών συνεργατικών σχηματισμών στον κλάδο του ICT, γιατί το ICT είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσο για τα πάντα, για τη γεωργία, για την ιατρική, για τα πάντα, ακόμα και για την αυτιλία. Έχουμε λοιπόν 10.000 μέλη που συνεργάζονται. Αυτά ξέρετε για την Ελλάδα κατά τα ε, χρόνια, τις δύσκολες περιόδους που διανύουμε, είναι ένα θαύμα. Και να σας πω ότι η ιδέα συνένωσης αυτών των ατόμων ήταν φανταστική γιατί πλέον συνεργάζονται, παράγουν, έχουν ε, συμμετοχές ε, και συμμετέχουν στην Silicon Valley σε ευρωπαϊκές, σε αμερικανικές εταιρείες οι οποίες έρχονται και παράγουν στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν βλέπετε ένα απλό παράδειγμα για δείκτες από την πρώτη στη δεύτερη φάση σε ό,τι αφορά ε, για παράδειγμα την ε, απασχολησιμότητα, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα. Όλοι αυτοί οι δείκτες έχουν διπλασιαστεί, μη σας πω και τριπλασιαστεί. Αυτό καταδεικνύει πόσο ε, όριμη είναι η κατάσταση. Βλέπετε λοιπόν τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται και τι προκύπτει από τη δεύτερη φάση από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, από την γοργή χρηματοδότηση 30 δισεκατομμυρίων και πλέον. 40 νέα προϊόντα έχουμε προωθήσει στην διεθνή αγορά. Το πρώτο που αναφέρεται είναι το MEMSense, ένα ε, project ε, πανεπιστημιακό, το οποίο είχε ε, εντυπωσιακά αποτελέσματα MEMSense σε ό,τι αφορά δίκτυα θητήρων. Έχουμε δύο κτίρια στην Αθήνα και στην Πάτρα. Ήταν ε, πραγματικά πολύ επιτυχημένο το εγχείρημα γιατί προσελκύει πραγματικά τους νέους που θέλουμε να τους κάνουμε επιχειρηματίες και από δίπλα είναι και τα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όπως είπατε και προηγουμένως. Το τρίτο ε, project ε, τονίζει τις νέους επιχειρηματίες και την επιτάχυνσή τους. Και θέτουμε ιδιαίτερη ε, έμφαση στα πανεπιστήμια. Και αυτό διαδίδει τις ιδέες των νέων. Κάθε χρόνο 20 άτομα στέλνουμε στο Stanford, στο MIT, στο Berkeley, στο Georgia Tech για να δουν τον Αμερικάνικο κόσμο. Έναν άλλον κόσμο, ο οποίος έχει εντάξει τους νέους στην αλυσίδα παραγωγής. Και φυσικά, ξεκινήσαμε με τη Eurobank. Αν το πιστεύετε, ε, μια τράπεζα ξεκίνησε το project EGG, EGG και πλέον έχουμε επιλέξει 23 επιχειρήσεις στο κτίριο μιας τράπεζας που δίνουμε συμβουλές και για ένα έτος θα έχουν σημαντικές ε, συμβουλές, θα λαμβάνουν σημαντικές συμβουλές, θα λαμβάνουν σημαντική καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τα θέματα επιχειρηματικότητας για το ελληνικό περιβάλλον. Είμαστε πλέον ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεργαζόμαστε για ευρωπαϊκά project για την ανάπτυξη της Νότια Ανατολικής Ευρώπης. Σε δύο project συμμετέχουμε. Το ένα είναι το ΕΝΕΚΟ, όπου το όραμα είναι να αυξηθεί η προώθηση, αν θέλετε, των κλάστερ, των συνεργατικών σχηματισμών στην Ευρώπη. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί. Εκπαιδεύουμε τους managers των κλάστερ, τους ε, τα διευθυντικά στελέχη των κλάστες σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό πηγαίνει πολύ καλά γιατί υπάρχουν μάνατζερ σε επίπεδο χωρών και οι κυβερνήσεις όλοι μαζί συνεργάζονται για την ανάπτυξη της χώρας προκειμένου να καταστούν πανευρωπαϊκοί φορείς και κλείνω στο σημείο αυτό να σας πω ότι το όραμα της πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς είναι η ανάπτυξη νέων στρατηγικών ε, για να ε, μεγιστοποιηθεί το δυναμικό επιχειρηματικότητας και προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική επιχειρηματική άποψη η συνεργασία. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει τη διαφορά, οι διεθνεί καλέ πρακτικέ, μια προσέγγιση από κάτω προ τα πάνω, έμφαση στην ε, καινοτομία και στην εξαγωγή, το ταλέντο, ο κόσμο πραγματικά ισχυρή η βιώσιμη μορφοποίηση των συνεργατικών σχηματισμών. Η Ελλάδα μας έχει υποβάλει προτάσεις για επιχειρηματικότητα, για επιχειρήσεις ε, στην περιοχή σε ό,τι αφορά την φορολογία, την ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση. Είμαστε σύμβουλος και της κυβέρνησης. Συμμετείχαμε στην ε, ανάλυση κινδύνου για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα κλάστερ και τη σχετική ανάπτυξη πολιτικής. Και αν θέλετε, το δυναμικό της Ελλάδας είναι η γεωργία, η ναυτιλία, ο τουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε την τεχνολογία ICT. Γιατί αυτό είναι το κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης σε οποιονδήποτε κλάδο. Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι απευθυνόμενος προς εσάς, προς την Ευρώπη, σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο καθεστώς και νομοθεσία για τις ευρωσυντεχνίες, μια ενιαία αγορά και αυτό λείπει για τα επιχειρηματικά κεφάλαια στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε και αυτό που αναφέρουμε ως ε, επιχειρηματικοί άγγελοι, ιδιώτες επενδυτές και όλα αυτά για να βελτιωθεί το clustering, για να βελτιωθεί η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φυσικά εντοπισμό των ευκαιριών για την καινοτομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ICT μπορεί να βοηθήσει και την γεωργία να δημιουργήσει, αν θέλετε, ε, πυρήνες ανάπτυξη στη χώρα, να εμπλέξει και να δώσει μια ευκαιρία και στους νέους να συμμετάσχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εσάς για, αυτή, την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Τώρα δίνω το λόγο στον δόκτωρο Όρταγα Αργυλές που ειδικεύεται στην εξειδίκευση. Έχετε το λόγο. Αν Και εσείς έχετε 10 λεπτά. Ε, hello, good morning. Ε, Γεια σας, καλημέρα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ ιδιαίτερος για την πρόσκληση. Είχα πολλές ιδέες για αυτή την παρουσίαση και έχω κάνει πολλές ε, παρουσιάσεις τα τελευταία τρία χρόνια για την ευφυή e e εξειδίκευση και εστίασα αυτήν εδώ στα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής βάσει των όσων γίνονται στις ε, χώρες του νότου της Ευρώπης. Σχηματικά θα σας παρουσιάσω το περιβάλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, το γνωρίζετε όλο. Θα σας παρουσιάσω τις αρχές της φιούς ε, εξειδίκευσης, εστιάζοντας τη βιομηχανία και μετά έχω διαμορφώσει διάφορες προκλήσεις για τον νότο της Ευρώπης που εμφανίζονται στις μελέτες περιπτώσεων για τις περιφέρειες και θα σας αναφέρω τις προκλήσεις αυτές που υπάρχουν για την υλοποίηση των στρατηγικών ευθείους εξειδίκευσης. Θα σας δείξω μια διαφάνεια με τα διάφορα βήματα που έχουμε συμπεριλάβει σε οδηγό που έχουμε δημοσιεύσει το 2010 για τις περιφέρειες και μετά θα περάσω κάποια παραδείγματα βάσει αυτών των μοτίβων επαναβιομηχάνησης, ε, όχι της υλοποίησης. Και τέλος θα σας δείξω πώς βάσει όλων αυτών των μελετών σε διάφορε περιφέρειες στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και κάτι μου λείπει ναι, και στην Πορτογαλία. Ποια είναι τα μοτίβα, ποιες είναι οι προτεραιότητες κατά τομέα που επέλεξαν μέχρι στιγμής. Όπως είπα λοιπόν, θα περάσω αυτή τη διαφάνεια. Ζητώ συγγνώμη που δεν έστειλα την παρουσίασή μου εκ των προτέρων. Αν κάποιο επιθυμεί να αποκτήσει το έγγραφο, μπορεί να μου το ζητήσει. Οι στρατηγικές εφηείους ε, εξειδίκευση ε, οι αρχές ε, για αυτή την περίπτωση των κλάστερ και της ανταγωνιστικότητας η κύρια είναι ότι δεν υπάρχει μία λύση κατάλληλη για όλους. Αυτές οι στρατηγικές λοιπόν εφίους εξειδίκευσης πρέπει να ε, είναι ενοποιημένες και να ακολουθούν μια προσέγγιση κατά τόπους, δηλαδή να εξετάζουμε σε ποιες περιφέρειες, σε ποιες περιοχές θα υλοποιηθούν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου περιβάλλοντος και της συγκεκριμένης κοινωνίας όπου θα υλοποιηθούν. Οι πολιτικές λοιπόν πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα μοτίβα βιομηχανοποίησης που υπάρχουν ήδη. Έχουμε δει διάφορες λοιπόν οδούς για την καινοτομία και την ανάπτυξη στις περιφέρειες, ε, ειδικότερα με βάση τη βιομηχανοποίηση, αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα. Ειδικότερα κάποιες περιφέρειες προσπαθούν να ανανεώσουν παραδοσιακούς τομείς με νέες τεχνολογίες, με διαφοροποίηση των τεχνολογιών με χρήση πολλών τεχνολογιών από διάφορους τομείς, με την ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω τεχνολογικών αλλαγών και καινοτομιών, όπως συμβαίνει στις Βαλεαρίδες, με τον τουρισμό, με νέες τεχνολογίες πληροφοριών υψηλής τεχνολογίας, αξιοποιώντας νέες ε, μορφές καινοτομίας, όπως την κοινωνική καινοτομία, όπως συμβαίνει στην Ιταλία με την ιστορική κληρονομιά. Ορισμένες από τις κοινέ προκλήσεις και πιθανές δράσεις που θα πρέπει να αναλυθούν σε αυτές τις περιφέρειες των χωρών του Νότου της Ευρώπης ε, μπορούν κάπως να ταξινομηθούν σε κοινωνικές ε, ουσιαστικά προκλήσεις. Έχουμε τεράστια προβλήματα ανεργίας σε πολλές περιοχές. Αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάρτιση, με αναβάθμιση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, ειδικότερα έχουμε υψηλή ανεργία των νέων που φτάνει στο 60% στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Επίσης έχουμε το πρόβλημα της γύρανσης του πληθυσμού. Αντί όμως να είναι αυτό πρόβλημα θα έπρεπε να αποτελεί ευκαιρία. Έχουμε διαπιστώσει λοιπόν ότι αναλαμβάνονται δραστηριότητε σε ορισμένε περιφέρειε, υλοποιούνται κάποια μέσα για να υλοποιηθούν οι νέε λύσει επιχειρηματικότητα ε, για να παρέχονται νέε υπηρεσίε όπω υπηρεσίε υγεία ή τρόπου ζωή διαβίωσης. Επίσης έχουμε και κάποια προβλήματα ε, συγκεκριμένα για συγκεκριμένους πληθυσμούς, ειδικότερα για τον πληθυσμό των ατόμων υψηλών ικανοτήτων. Χρειάστηκε λοιπόν αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων και των ερευνητών. Χρειάστηκε βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, της προσβασιμότητας και της προσέλκυσης. Επίσης διαπιστώσαμε πολλά προβλήματα αποφυγής των κινδύνων, δηλαδή η επιχειρηματική κουλτούρα δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Ενθαρρύνουμε λοιπόν δραστηριότητες προώθησης της επιχειρηματικότητας και στην εκπαίδευση στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στη δευτεροβάθμια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις σχετικές δραστηριότητες και έχουμε διαπιστώσει ότι σε πολλές περιφέρειες υπάρχει δυσπιστία ε, ως προς ε, τα κρατικά όργανα και μια διαρκής θεώρηση ότι οποιαδήποτε περιφερειακή στρατηγική μπορεί να τους εξυπηρετήσει ως ε, προς το γεγονός ότι αποκτούν η οικειοποίηση, η ιδιοκτησία αυτής της στρατηγικής. Υπάρχουν και κάποιες προκλήσεις για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης. Υπάρχει το πρόβλημα της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης, οποιαδήποτε βελτίωση των δραστηριοτήτων σε κλάστερ, ακόμη και τα μοτίβα επανεκβιομηχάνησης δεν πρέπει να βασίζονται μόνο σε κονδύλια που λαμβάνονται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτά πρέπει, πρέπει να υπάρχει και ε, μια συμπληρωματική χρηματοδότηση από διάφορες πηγές. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιφέρειες. Υπάρχει ένα διπτό πρόβλημα. Χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και στο φυσικό κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα λόγω της ύφεση υπάρχουν και χαμηλές δημόσιες επενδύσεις. Προβλήματα λοιπόν πρόσβασης σε ρευστό. Πιθανώς λοιπόν σε κάποιες από αυτές τις χώρες η πρόκληση αναλογικότητα όσον αφορά την υλοποίηση του κινδύνου είναι υψηλότερη από τις άλλες χώρες. Επίσης υπάρχει τεράστιος κατακαιρματισμός και περιτές εργασίες. Το ξαναείδαμε. Οι περισσότεροι τομείς ε, που προωθούνται είναι σχεδόν οι ίδιες δραστηριότητες, σχεδόν οι ίδιοι υποτομείς σε πολλές περιφέρειες. Πρέπει να αποφεύγεται αυτός ο διπλασιασμός πρέπει να δούμε σε ποιο σημείο έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια συγκεκριμένη περιφέρεια ώστε να του συστήσουμε πιθανές συνεργασίες με άλλες περιφέρειες ε, σε άλλες χώρες μέσω διαφορετικών εταιριών στην Ευρώπη. Επίση υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα του ownership, της οικειοποίησης. Έχουμε ισχυρά μοτίβα εξασκής σε ορισμένες περιφέρειες και αυτό αποθαρρύνει την ιδιωτική συμμετοχή, την εμπλοκή των ενδιαφερομένων, διότι γνωρίζουν σε ορισμένε περιπτώσει ότι πάντα οι ίδιε επιχειρήσει είναι εκείνες που λαμβάνουν επιχορηγήσει και τα παρόμοια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια διαδικασία διαβούλευση με του ενδιαφερόμενου, ώστε να του δείξουμε ότι η οικειοποίηση, τα ωφέλη των στρατηγικών που θα υλοποιηθούν θα κατανεμηθούν ε, ισότιμα μέσω όλων των συμμετεχόντων στη στρατηγική έχουμε, διότι στις συγκεκριμένες αυτές χώρες υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ περιφερειών. Υπάρχουν λοιπόν και προβλήματα σε ορισμένες από τις χώρες προσβασιμότητας, όπως στην Νότια Ιταλία. Επίσης πολλά προβλήματα λόγω της κλιματικής ε, αλλαγής, ε, όσον αφορά ας πούμε, τις διαδικασίες πιστοποίησης ε, στις νότιες χώρες, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και αυτές οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία ανάδυσης νέων βιομηχανιών όπως η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση των αποβλήτων, η ανακύκλωση των αποβλήτων σε ορισμένα νησιά. Αρχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των τομέων εκβιομηχανήσης που θα πρέπει να προωθηθούν και τέλος οι προκλήσεις καινοτομίας και τεχνολογίες είναι κατακαιρματισμένες και ε, περιορίζονται λόγω των κανονισμών που υπάρχουν, των ρυθμίσεων που υπάρχουν για την καινοτομία και τις ε, επιστήμες. Επίσης χαμηλή αποτελεσματικότητα μετατροπής της ε, έρευνας σε καινοτομία. Αυτό που αναφέρατε, ότι, που έρευνε ο Πορτογάλος συνάδελφος εδώ, ότι θα μπορούσε να προσθέσει αξία. Αυτά είναι τα βήματα που ορίζει ο οδηγό για να διευκολύνει τι περιφερειε να προχωρήσουν προ τα εμπρό για να επινοήσουν νέε στρατηγικέ. Δεν θα σα τα παρουσιάσω λεπτομερώς, πιστεύω ότι τα γνωρίζετε όλοι, αλλά θα χρησιμοποιήσω κάποια από τα βήματα για να σα δώσω κάποια παραδείγματα. Στο πρώτο βήμα, στην ανάλυση, εκεί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα προφίλ τη περιφέρειας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκεί έχουμε και τις διαφορές ε, συνθήκες των διαρθρωτικών ταμείων. Ψάχνουν για μια ανάλυση, ότι προσπαθούν να βρουν τα ισχυρά σημεία, τα δύναμα σημεία, τις ευκαιρίες που έχει μια περιφέρεια. Πέραν αυτή της ανάλυσης έχουμε δει ότι σε κάποιες περιφέρειες συμπληρώνουν αυτή την ανάλυση με ανάλυση οροσίμων ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστικούν παγκοσμίω. Έχουν λοιπόν οριοθετήσει ορόσημα και σε συνεργασία με γειτονικέ περιφέρειε ε, εντό των κρατών μελών και διεθνώ. Ένα παράδειγμα στην Ισπανία είναι το παράδειγμα τη Ναβάρα που αναζητά ώστε να βρει σε παρόμοιες περιφέρειες ε, αντίστοιχες περιπτώσεις ώστε να μην διπλασιάζονται οι εργασίες. Πριν θέσουν προτεραιότητες ε, αναζητούν τι δυνατότητες συνεργασίας στο θέμα της διακυβέρνησης και της δημόσιας διαβούλευσης, πολλές ε, περιφέρειες προσπαθούν να εμπλέξουν ε, όσο περισσότερο δυνατό τους ενδιαφερόμενους. Θα περάσω τώρα στις προτεραιότητες. Εδώ βλέπουμε πώς ε, προσπαθούν να βρουν τα μοτίβα επανεκβιομηχάνηση που πρέπει να ακολουθήσουν στην περίπτωση της Ναβάρα στην Ισπανία οι στρατηγικοί κλάστερ που ακολουθούν ότι προσπαθούν να αναπτύξουν διάφορα κλάστερ ανάλογα με τη σπουδαιότητα που έχουν οι συγκεκριμένοι τύποι βιομηχανιών για την περιοχή της Ναβάρα, δηλαδή κλάστερ συγκεκριμένα διατήρησης της απασχόλησης στα επίπεδα στόχους ή στρατηγικές που βοηθούν να παρασχεθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα οι τομεί όπου έχει σημαντική παρουσία η Ναβάρα ή συμπληρωματικέ πτυχέ όπω η εκπαίδευση. Στην περίπτωση τη Εμίλια Ρωμάνια στην Ιταλία, είδαν τι προκλήσει κλειδιά. Είναι δύο. Η μία είναι αναβάθμιση των παραδοσιακών τομέων και η άλλη είναι η ενίσχυση των αναδυόμενων κλάστερ. Ακολούθησαν λοιπόν κάποια κριτήρια για να αναλύσουν το ποιες δραστηριότητες θα ακολουθήσουν. Έχουμε διαμορφώσει πολλά έτσι, παραδείγματα, μπορείτε να δείτε σε αυτή τη διαφάνεια και πολλές αναλύσεις. Τώρα όσον αφορά την υλοποίηση σας δίνω κάποια παραδείγματα των διαφόρων δυνατοτήτων τι θα μπορούσε να ακολουθήσει κανείς ώστε να υλοποιήσει ένα μείγμα πολιτικών που θα υποστηρίξει αυτή την ανάλυση κλάστερ όπως ε, ελκυστικότητα των βιομηχανιών, κίνητρα για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και της ε, μεταφοράς τεχνολογιών με θεματικές πλατφόρμες, με περιφερειακά δίκτυα, αναβάθμιση τεχνολογική με συγκεκριμένη τεχνική εκπαίδευση και ορισμένα παραδείγματα μπορούμε να δούμε στην περίπτωση της Καστίγια Λαμάντσα στην Ισπανία όπου δημιουργείται ένα σύστημα ανάπτυξης voucher γνώσης όπου δαπανώνται χρήματα σε περιφερειακά πανεπιστήμια για να διευκολυνθεί το να μάθουν αυτά τα περιφερειακά πανεπιστήμια πώς να συνεργάζονται για να γίνουν οι τοπικές επιχειρήσεις παγκόσμια πιο ανταγωνιστικές. Σε περίπτωση που δεν έχουν υπάρξει συνεργασίες με τις επιχειρήσεις είναι αδύνατη αυτή η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Και εδώ έχουμε και άλλο ένα παράδειγμα και μετά από αυτό θα ολοκληρώσω. Δεν είναι νότια χώρα της Ευρώπης, είναι στις κατοχώρες, η επαρχία του Λιμβούργου, μια μακροπεριφέρεια που δημιουργήθηκε με 19 περιφέρειες που ανήκουν σε 4 χώρες στο κέντρο της Ευρώπης και εκεί προσπάθησαν να δημιουργήσουν αυτή την κρίσιμη μάζα αλλά επειδή ενίοτε έχουν τη βασική έρευνα, έχουν τα πανεπιστήμια, αλλά δεν έχουν τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται στις έρευνες που διεξάγουν αυτά τα πανεπιστήμια. Και έχουν και πολλούς εργαζομένους που ταξιδεύουν για τη δουλειά τους, για να πάνε στη δουλειά τους. Και το καλύτερο μοτίβο ήταν να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των περιφερειών που ανήκουν σε διαφορετικές χώρες. Και εγώ παρέχοντα συμβουλέ στι χώρε του Νότου, του ζητώ να παρατηρούν και τι γίνεται όχι μόνο στι δικέ του χώρε, αλλά και τριγύρω σε άλλε χώρε. Αυτά εδώ είναι τα μοτίβα που διαπιστώνουμε σήμερα, τα μοτίβα επανακβιμηχάνησης, μελετώντας τις μελέτες περιπτώσεων όλων αυτών των περιφερειών μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ζητώ συγγνώμη που κάποιες στιγμές χρειάζεται να σας διακόψω και που σας πιέζω με το χρόνο, αλλά πώς να το κάνουμε ο χρόνος σήμερα είναι δυστυχώς περιορισμένος και θέλω να αφήσω περιθώριο και για τη συζήτηση, τη συζήτηση στην οποία έχουν γραφεί ήδη κάποιοι συνάδελφοι. Υπάρχουν δύο λεπτά για τον κάθε ομιλητή για να κάνετε τις ερωτήσεις σας, ώστε οι ομιλητές μας να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν. Τον κύριο Μπιτικόφερ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σιγητή αν θέλει να παρέμβει και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι μία ερώτηση προς τον Έλληνα εκπρόσωπο σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να παίζουν οι, οι επιστήμονες που βρίσκονται σε άλλες χώρες σε σχέση με την προώθηση των clusters. Είδαμε ότι οι εκπατρισθέντες Ινδοί και Κινέζοι έπαιξαν ένα σημαντικότατο ρόλο στο Silicon Valley και βοήθησε αυτό να προκόψουν και οι χώρες τους η Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο δεν αντιμετωπίζει επιτυχώς την λεγόμενη φυγή των εγκεφάλων από τις ευρωπαϊκές χώρες. Μήπως μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη, να μην μιλάμε για brain drain, αλλά να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε ε, την επιτυχία και τις ικανότητες των ομογενών σαν παράδειγμα που βρίσκονται σε άλλες χώρες και έχουν πετύχει εκεί. Κοιτάξτε, θα ακουστούν όλες οι ερωτήσεις και μετά θα μας απαντήσετε. Η Πιλάρντε Καστίλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τους δύο προηγούμενους ομιλητές, όποιος θέλει μπορεί να σχολιάσει να απαντήσει. Αφορά το ICT. Το ICT στην πραγματικότητα είναι ένας οριζόντιος πλέον παράγων. Ε, θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να διαπεράσει το σύνολο της κοινωνίας και των βιομηχανιών. Ως εκ τούτου λοιπόν, καλό θα είναι να ασχοληθούμε με αυτό με πιο εξειδικευμένο τρόπο. Όταν μιλάμε για τα ICT, για την έλλειψη, την ανάγκη που μπορεί να έχουμε, είναι απαραίτητο σε μερικές περιπτώσεις να επαναπροσανατολίσουμε τις αναλύσεις μας και τις προσπάθειες έβρεσης διαγνώσεων για το τι χρειάζεται ο Νότος, τι χρειάζεται το κέντρο της Ευρώπης και ε, ο βοράς της Ευρώπης από το επίπεδο το πανεπιστημιακό μέχρι το επίπεδο της παραγωγής μέχρι το επίπεδο των υποδομών γιατί τώρα μιλάμε για τεράστιες ανάγκες στη μεταφορά δεδομένων, κάτι το οποίο θα βοηθήσει επίσης να ασφαλίσουμε τα δίκτυά μας και να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη σε αυτά. Εσείς πώς βλέπετε η Ευρώπη να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα στο νότο της Ευρώπης. Τι ρόλο παίζουμε. Γιώχανσον. Ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές για τα ξεκάθαρα μηνύματα τα οποία μας μεταφέρατε. Πριν γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήμουν περιφερειακός υπουργός σε μία από τις ε, βιομηχανικές περιοχές της ε, Σουηδίας και τα περιφερειακά κλάστερ είναι πολύ σημαντικά αρκεί να είναι ανοιχτά στην παγκοσμιοποίηση. Εδώ έχουμε πολλά κοινά με τα περιφερειακά επίπεδα που ισχύουν γενικότερα στην Ευρώπη. Δυστυχώς βέβαια πολλές φορές σε εθνικό επίπεδο οι αντιλήψεις είναι διαφορετικές. Εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε τις ιδέες αυτές ε, των κλάστερς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βιομηχανία ε, είναι θέμα όμως το οποίο θα πρέπει να τεθεί προσυζήτηση και στο Συμβούλιο και αν πράγματι ακολουθήσουμε αυτά τα μηνύματα τα οποία εσείς μας μεταφέρατε, τι γίνεται με τον ανταγωνισμό. Και αν χρησιμοποιούμε την λέξη Ευρώπη, το επίθετο ευρωπαϊκός, αυτό τι ρόλο μπορεί να παίξει σε επίπεδο κρατών μελών. για την δημιουργία περιφερειακών κλάστερς ανοιχτών όμως στον υπόλοιπο κόσμο. Πολλές φορές οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες αυτές σε εθνικό επίπεδο είναι λίγο ε, εσωστρεφείς θα έλεγα και μερικές φορές και ο λίγο υπερπροστατευτικοί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε λίγο τι σκέφτεστε για το τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο φυσικά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά με ενδιαφέρει το επίπεδο των κρατών σε αυτή τη φάση. Ο πρώτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές γιατί πράγματι τα μηνύματά τους και τα ρεθίσματά τους ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Θα ήθελα λίγο να προσπαθήσουμε να δούμε τι λάθη έχουμε κάνει στο παρελθόν και πώς αυτά τα λάθη φωτίζονται σήμερα και πώς θα τα καταλάβουμε σήμερα. Καταρχάς, εμείς θεωρήσαμε τη μεταποιητική βιομηχανία σαν χαμένη πια, την ξεχάσαμε. Είπαμε την αγγλική φράση «It's globalization stupid» και τα ξεχάσαμε όλα τα άλλα. Ενώ υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες είχαν τον πολιτισμό της προσαρμογής και της παραγωγής στον τομέα τον μεταποιητικό και είχαν επίσης και τις επαφές και την επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις και με άλλες περιοχές του κόσμου. Εδώ λοιπόν είναι προφανής η έλλειψη μια ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής και καινοτόμου βιομηχανικής πολιτικής. Και εδώ έρχεται και κάτι άλλο να επιβαρύνει την κατάσταση. Εμείς αξιολογήσαμε τις επιχειρήσεις αποκλειστικά από το μέσο του παράγοντα της παραγωγικότητας. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν αποκλειστικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας επιχείρησης θα πρέπει να κατανοήσουμε την αξία μιας επιχείρησης και μέσω από τις θέσεις εργασίας και μέσω του πολιτισμού που προσφέρει σε μια περιοχή. Αναφέρομαι σαν παράδειγμα ε, στο κλάστερ συσκευασιών που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια στην Ιταλία. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ και έχει την ικανότητα το κλάστερ αυτό να δημιουργήσει ένα supply chain, μια οργάνωση εδαφική γύρω από την παραγωγή της. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενισχύει αυτές τις βιομηχανικές περιοχές μέσω των κλάστερς και προσδίδει σε αυτές τις βιομηχανικές περιοχές μία διεθνή, μία παγκόσμια διάσταση διατηρώντας την ανεξαρτησία των περιοχών αυτών και διατηρώντας ζωντανό το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Από αυτό λοιπόν πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Θα πρέπει να βλέπουμε φυσικά τα καλά παραδείγματα των startups αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να μην ξεχνάμε το σύνολο παραγωγικού δίκτυο μιας περιοχής το οποίο έχει λειτουργήσει και θα πρέπει εξ αρχής να αξιολογούμε σωστά τις επιχειρήσεις και για την άειλη σημασία τους, την οργανωτική, πολιτισμική ε, ε, συνεισφορά τους στην μεταποιητική δραστηριότητα γενικά. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους εμπειρογνώμονες, τους οποίους ευχαριστώ και εγώ. Η τρίτη παρουσίαση ε, θα μας την αφήσει η Ισπανίδα συνάδελφος γιατί δεν την έχουμε. Τις άλλες τις έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω ποιος θα αρχίσει τις απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, expats, των εκπατρισμένων, να σα πω ότι θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ένα ταλέντο σε όλο τον κόσμο δυσπαρμένο, πραγματικά υπέρ της αξίας. Εγώ ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχω στείλει πάνω από χιλιά άτομα στο εξωτερικό και θέλω να επιστρέψουν. Το 99 φέραμε μια αμερικανική εταιρεία με Έλληνες ιδιοκτήτες την ADMIL στην Πάτρα και έτσι ξεκίνησε ένα κλάστερ μικροηλεκτρονικής. Η ιδέα λοιπόν ήταν οι Έλληνες του εξωτερικού να δράσουν ως γέφυρα και να δημιουργήσουν ε, κέντρα design σχεδιασμού για νέα ανάπτυξη ICT. Αυτό μπορεί να συμβεί και με ευρωπαϊκές εταιρείες που δεν έχουν όχι με κόσμο που φεύγει από την Ελλάδα και πάει στην ε, Γερμανία, αλλά δημιουργώντας θηγατρικές επιτόπου και έτσι χρησιμοποιώντας τον κόσμο αυτό, αξιοποιώντας τα δυνατότητες του κόσμου αυτού, ο οποίος εργάζεται πλέον στον τόπο του και αυτό δεν η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Να σας πω ότι στην ε, Ελλάδα, στην ηλεκτρονική μηχανική, στη βιοτεχνολογία έχουμε το πιο υψηλό επίπεδο ε, εξετάσεων ε, εισαγωγής. Αλλά δεν μπορεί να βρει δουλειά αυτός ο κόσμος και γι' αυτό λοιπόν το clustering είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δημιουργούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για να χρησιμοποιηθούν, να αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν είναι το καθήκον, ο σκοπός του Κοράλια. Στο θέμα τα παγκοσμιοποίησης να σας πω ότι τα κλάστερ σε μικροελεκτρονικής το να είναι, το κλάστερ όριμο και για τα επίπεδα της Ελλάδας αλλά και για τα επίπεδα του εξωτερικού. Μιλάω για κάτι πρόσφατο. Με 78.000 ε, άτομα στην ε, Silicon Saxony, στην Grenoble έχουμε 50.000 άτομα, DSP στο Βέλγιο, NXP στην Ολλανδία, Μόντσα στην Ιταλία. Με όλα αυτά λοιπόν δημιουργούμε ένα κλάστερ παγκόσμιου βεληνικούς. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος προς τα εμπρός και το clustering θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο τα τελευταία 15 χρόνια. Μπορεί λοιπόν να δημιουργήσει αυτή την προσέγγιση παγκοσμιοποίησης. Για να απαντήσω στο ερώτημά σα. θα πρέπει να σκεφτούμε εκ νέου πώς θα διαμορφωθεί η βιομηχανία και αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος ο μοναδικός τρόπο να, το, να επαναεφεύρουμε την βιομηχανία είναι να σκεφτούμε τι έγινε στο Silicon Valley, τα μεγάλα πανεπιστήμια, ε, Stanford και ούτω καθεξής. Πήγε λοιπόν η Silicon Valley στα πανεπιστήμια αυτά και είπε πείτε μας ποια ήταν η ιδέα αυτού του λαμπρού μυαλού. Ας αναπτύξουμε την ιδέα αυτή. Στην ε, Ευρώπη τα μεγάλα πανεπιστήμια, και δεν θέλω να τα κατανομάσω, θα πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν πώς οι μεγάλε ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε καινοτομία. Και γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε την τεχνολογία ICT, γιατί τα συστήματα ε, σε ό,τι αφορά τα chips, τα embedded systems, μπορούν να αλλάξουν την ιατρική, την γεωργία, τον τουρισμό. Αναδεικνύοντα τουριστικά project, για παράδειγμα στη δήλωση στην Ελλάδα, α πούμε, να αναφέρουμε ότι μιλάμε για την πιο καλά διατηρημένη αρχαία πόλη στην, ε, στον κόσμο. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν ένα project για να ε, δημιουργηθεί και να αναδομηθεί η δήλωση με την τεχνολογία Avatar. Αυτό. Και τήρησα και το χρονοδιάγραμμα, κυρία Πρόεδρε. Λίγο πολύ απαντάει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που θέσατε. Εγώ ήμουν εμπειρογνώμων σύμβουλο στην Εκτρεμαδούρα, στην Καστία Λαμάντσα, στην Ισπανία και συνεχίζω να αξιολογώ το έργο τους εκεί όσον αφορά την υλοποίηση τη έξυπνης ε, εξειδίκευσης και ειδικότερα σε περιφερειές σαν αυτή έχουν τεράστιο πρόβλημα δεξιοτήτων, ικανοτήτων για να προσελκύσουν ανθρώπους από, και ε, μάλλον πολυεθνικές για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ε, το πρόβλημα είναι το να υπάρξει το κατάλληλο περιβάλλον, ο εξυγχρονισμός, ώστε αυτές οι πολυεθνικές να θέλουν να πάνε σε τέτοιες περιφέρειες. για αυτό το σκοπό έχουν ένα εξαιρετικό τμήμα στα πανεπιστήμια ε, Φωτονική στην Καστίγια Λαμάντσα, άριστης ποιότητας, ανταγωνίζεται παγκοσμίω. Συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, αλλά κανείς σε τοπικό επίπεδο δεν έχει καμία σχέση με αυτού του είδους τα τμήματα. Και εγώ μια φορά σε μια συνέντευξη με τον διευθυντή μου είπα ότι είναι απόλυτο διατεθειμένοι να συνεργαστούν με τη βιομηχανία σε τοπικό επίπεδο για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, για την ηλιακή ενέργεια και όλα τα σχετικά. Αλλά φυσικά οι επιχειρήσεις της περιφέρειας, στην Καστίγια Λαμάντσα ή στην Εξτρεμαδούρα που επίση θέλουν να δώσουν προτεραιότητα σε αυτού του είδου ενέργειε δεν γνωρίζουν τίποτα για την έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό το σκοπό προσπαθώ να προωθήσω περισσότερο αυτά τα knowledge vouchers περιφερειακά ή τοπικά ώστε να ενθαρρυνθεί αυτή η συνεργασία, ώστε οι επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά σε πανεπιστήμια σε αυτές τις συγκεκριμένες περιφέρειες να ενθαρρυνθει αυτη η συνεργασια ωστε οι επιχειρησεις που βρισκονται κοντα σε πανεπιστημια σε αυτέ τι συγκεκριμένε περιφερειες να γνωριζουν τι έρευνε διεξάγονται στα πανεπιστήμια των συγκεκριμένων περιφερειών και έτσι να μπορέσει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πανεπιστημίων. Αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η δημιουργία διεξιοτήτων, ανθρώπων, ανθρώπινου δυναμικού που να έχει τις δεξιότητες ώστε να μπορέσει να προσελκύσει οποιοδήποτε τύπο βιομηχανία. Διαφορετικά ε, χάνουν διαρκώς κρίσιμη μάζα, την οποία χρειάζονται. Ένα άλλο θέμα για την παγκοσμιοποίηση είναι η διαδικασία ενημέρωσης πρέπει να ενημερώνουν για το τι μπορούν να κάνουν καλά, πού μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Όλοι θέλουν να κάνουν αγροδιατροφή, είναι εξαίρετοι, στη Γεωργία έχουν ειδικευμένα τμήματα αγροτικών μηχανικών, έχουν αναπτύξει καλλιέργειες και όλα αυτά, αλλά δεν συνεργάζονται. Και πάλι Συχνά αυτά τα πανεπιστημιακά τμήματα είναι γνωστά παγκόσμια λόγω διασκέψεων διεθνών και μεγάλε πολυεθνικέ πάνε σε τέτοιε διασκέψει και γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοιε δραστηριότητε στην Ευρώπη, αλλά τοπικά δεν γνωρίζει κανεί τι συμβαίνει εκεί πέρα. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ δυνα... σημαντικό μεν παγκοσμίω, αλλά είναι σημαντικό και τοπικά να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά το εθνικό επίπεδο, έχω δει πρωτοβουλίες. Πήγα στην Ιταλία και εκεί είχα μια συνάντηση με τον Φαμπρίζιο Βάρκα με πολλούς εκπροσώπους των Ιταλικών περιφερειών. Τι προσπαθούν να κάνουν εκεί. Προσπαθούν να παρακολουθούν την όλη διαδικασία υλοποίησης των στρατηγικών ευθείους εξειδίκευσης στις διάφορες περιφέρειες, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να διαμορφώσουν ε, τεχνολογικά μοτίβα, μια τεχνολογική χαρτογράφηση και προσπαθούν ε, να ορίσουν τις θέσεις ορισμένων περιφερειών σε αυτή τη χαρτογράφηση. Τι προσπαθούν λοιπόν να κάνουν, να ε, χρησιμοποιήσουν μια κοινή βάση ώστε να δημιουργήσουν αυτά τα κλάστερ σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Επειδή ταυτόχρονα διεξάγουν τις δύο αναλύσεις, εθνική και περιφερειακή. Υποστηρίζω λοιπόν τη συνεργασία του εθνικού και του περιφερειακού επίπεδου, αποδεικνύει την χρησιμότητα της συμπληρωματικότητας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ όλους μας τους φιλοξενούμενους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ας συνεχίσουμε τώρα. Συνεχίσουμε με το δεύτερο πάνελ που αφορά την αηφόρο επανεκβιομηχάνηση. Η πρώτη ομιλία θα είναι του Τζουζέπε Μπράτα, πρόεδρος ε, της, περιφέρειας, της παραγωγικής περιφέρειας της Απουλίας για τις ανανεώσιμες ενέργειες και την ενεργειακή απόδοση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η ομιλία μου θα επικεντρωθεί στον κόσμο της παραγωγής που διαρκώς δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής. Εγώ είμαι πρόεδρος της παραγωγικής ε, περιφέρειας της Απούλιας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια Ιταλική αριστεία θα έλεγα, στην Νότια Ιταλία, στην Απούλια. Θα σας διηγηθώ τις εμπειρίες μας από την περιφέρειά μας όταν στο 2010 αποφάσισε η περιφέρεια της απουλίας να νομοθετήσει περιφερειακά δημιουργώντας ένα μέσο συγκέντρωσης επιχειρήσεων παραγωγικών και δημοσίων αρχών που άρχισαν να συνεργάζονται σε αυτόν τον τομέα που έδειξε επιρροχή. Στο μέσο αυτό συμμετέχουν σήμερα 350 επιχειρήσεις, 13 τοπικές αρχές και όλα τα ερευνητικά, παρεπιστημιακά, δημόσια και ιδιωτικά κέντρα. Οι οργανισμοί αυτοί αντιστοιχούν σε 10.000 μέλη σε αυτόν τον τομέα που γεννήθηκε στην Απουλία πριν από 5 χρόνια ε, συνολικού προπολογισμού ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι επιχειρήσεις ανανόσμων πηγών ενέργειας ε, ασχολούνται με πολλούς διαφορετικούς τομείς, τον κλασικό τομέα της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αιωλικά, βιομάζα και τα λοιπά, ηλιακή ενέργεια, τις νέες πράσινες τεχνολογίες. Θα σας μιλήσω στο τέλος και για όλο το κομμάτι του φωτισμού και της ενεργειακής απόδοσης. Πριν μπω σε συγκεκριμένα νούμερα και σε συγκεκριμένες σκέψεις. ώστε να καταλήξω σε πολύ ευφυείς ε, συγκεκριμένες προτάσεις, θα ήθελα να σας παρουσιάσω μερικές γενικές σκέψεις. Αυτή τη στιγμή το παραγωγικό σύστημα της Ιταλίας και στην Απούλια ε, αποτελείται κατά 90% από μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ήδη έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι η καινοτομία και η, πτυχή, η περιβαλλοντική πτυχή αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την ίδια την ανάπτυξη, την αηφόρια και την μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται κάποιο είδους οδικό χάρτη, μια οδό που θα ακολουθήσουν μια λογική, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Τα κρίσιμα αυτά εδώ χρόνια οφείλονται στην έλλειψη οράματος μακροπρόθεσμου ουσιαστικά. Για να σας δώσω μερικά νούμερα, το 2011 το 75% της ιταλικής παραγωγής ενέργειας προερχόταν από ορυκτά καύσιμα ή από εισαγωγές το 25% από ανανεώσιμες πηγές. Η Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική, που ακόμα βρίσκεται υπό συζήτηση, προβλέπει ότι το 2020 το 62% θα αντιστοιχεί σε ορεκτές πηγές ενέργειας και το 38% σε ανανεώσιμες πηγές. Αυτό οδηγεί σε δύο σκέψεις. Το πρώτο είναι ότι το 2020 στο τομέα της ενέργειας ε, το 2020 για το τομέα της ενέργειας δεν απέχει πολύ. Χρειάζεται ίσως ε, μια μεγαλύτερη προθεσμία από 7 χρόνια. Ο σχεδιασμός σε αυτό το τομέα σημαίνει ότι χρειάζεται σχεδιασμός για τουλάχιστον άλλα 15 χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν σχεδιασμός τουλάχιστον μέχρι το 2030 με τα σημερινά μέσα που έχουμε αυτό το 38% στην Ιταλία πιθανώς δεν θα επιτευχθεί προβλε... όπως προβλέπεται από μελέτες της ηλεκτρικής, ε, Ιταλικής ηλεκτρικής αρχής ότι το πιθανότερο είναι με τις τρέχουσες, με το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο να φτάσουμε το 33%. Από το 2004 μέχρι το 2011 στην Ιταλία και στην Πούλια αναπτύχθηκε ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 65%. 75% στην πόλια. Περισσότερο δηλαδή δεκαπλάσιο σε σχέση με τον εθνικό μεσόρο. Η Απούλια αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη περιφέρεια της Ιταλίας στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς διατηρήσαμε αυτή την πρώτη θέση δίνοντας προτεραιότητα στις μεγάλες εγκαταστάσεις ε, από οικονομική άποψη, στις εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά. Η Απούλια στον τομέα των φωτοβολταϊκών είναι η πρώτη περιφέρεια από άποψη παραγωγής, αλλά όχι η πρώτη από άποψη πλήθους εγκαταστάσεων. Αυτό μας αποδεικνύει ότι μέχρι στιγμής στην Απούλια έχουν αναπτυχθεί μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εγκαταστάσεις που υλοποιήθηκαν στην παρούσα φάση στις αγροτικές περιοχές, σε αγροτικά εδάφη. Αυτή η πρώτη φάση είναι μια φάση που έχει ολοκληρωθεί. Μια δεύτερη φάση τώρα θα βασίσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ιδέα της αηφορίας του εδάφους. Στην ιδέα της του εδάφους αηφορία σε, βασισμένη σε εδάφη μικρού μεσαίου μεγέθους που θα βασιστούν στην αυτοκατανάλωση, δηλαδή εγκαταστάσεις μικρού μεγέθους, μήνυα ολικές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν αγροκτήματα και, και μικρές εγκαταστάσεις βιομάζας. Κάποια στοιχεία για τις επιπτώσεις της green economy στην ε, εργασία. Πολλές μελέτες έχουν δείξει αντικειμενικά ότι οι επιπτώσεις ε, της green economy στις θέσεις εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντικές, ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά έχουν οκταπλάσια ε, ε, αποτελέσματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής ενέργειας. 10.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην Απούλια. Αυτά τα 10.000 άτομα που εργάζονται καθημερινά είναι όλοι νέοι κάτω των 40 ετών όλοι νέοι επαγγελματίες. Μιλάμε δηλαδή για νέους μηχανικούς, τεχνικούς, ε, επαγγελματίες που πιστεύουν σε αυτόν τον τομέα και θέλουν να συνεχίσουν να πιστεύουν σε αυτόν. Eh, σε αυτή την ανάπτυξη που έλαβε χώρα σε αυτό το τομέα στην Παπούλια, σίγουρα Γι' αυτό τον τομέα ακούστηκαν και πολλές κριτικές. Και κάποια, έγιναν σίγουρα και κάποια ασφάλματα, διότι αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτη κριτική, η αβεβαιότητα του κανονιστικού πλαισίου. Να σας δώσω ένα στοιχείο, τα τελευταία τρία χρόνια οι επιχειρήσεις που επένδυσαν σε αυτό τον τομέα είδαν να αλλάζουν οι κανόνες τρεις φορές. Δηλαδή κατά μέσο όρο μία φορά το χρόνο. και πολλές φορές μέσα στον ίδιο χρόνο άλλαζαν πολλά πράγματα ή υιοθετούν τα πράγματα με τρίμηνης ισχύω ε, το οικονομικό σύστημα σήμερα δεν ε, μπορεί να καλύψει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικότερα των βιώσιμων μορφών ενέργειας. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της μεγαλύτερης Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κονφάμπη που απαριθμεί 120.000 επιχειρήσεις μικρομεσαίες στην Ιταλία έδειξε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλουν αόριστα κίνητρα, θέλουν απλά ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να έχουν σταθερότητα μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι το αίτημα. Η ευχή όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η γραφειοκρατία είναι το κυριότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη αυτού του τομέα. Δυστυχώς στην Ιταλία για να κατασκευάσει κανείς ε, μια εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρειάζεται περίπου 30 άδειες. Είναι αδύνατο να υπάρξει ανάπτυξη όταν η γραφειοκρατία είναι τόσο μεγάλη. Μια άλλη τεχνική πτυχή, λειτουργική πτυχή είναι η έλλειψη δικτύων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας δεν μπορούν να κατασκευαστούν πλέον εγκαταστάσεις, εργοστάσια, διότι οι υποδομές, τα δίκτυα μεταφοράς δεν είναι επαρκή. Στην πρώτη φάση, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, δόθηκε προτεραιότητα σε οικονομικές επενδύσεις. Σε μια δεύτερη φάση θα δοθεί προτεραιότητα σίγουρα σε διαρθρωτικές επενδύσεις. Προτάσεις smart τώρα για την ανάπτυξη, το να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πρόθεση και στην καινοτομία, το να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε όλη τη γραφειοκρατία, ευχόμενη να υπάρχει ίδια γραφειοκρατία σε όλη την Ευρώπη να προσδιοριστούν τα κίνητρα και τα φορολογικά κίνητρα που θα είναι μοναδικά σε όλη την Ευρώπη και μια πρόταση που θα πρέπει να προωθηθεί κατά την άποψή μας είναι ότι η ανάπτυξη αυτού του τομέα πρέπει να λαμβάνει η χώρα σε όλους τους τόπους όπου καταναλώνεται ενέργεια. Δηλαδή ευχόμαστε κάθε καταναλωτής, κάθε επιχείρηση να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται. Για αυτό δεν χρειάζονται μεγάλοι πόροι. Χρειάζεται βεβαιότητα από αψή γραφειοκρατίας. Κάθε επιχείρηση πρέπει να μπορεί να παράγει την ενέργεια που της χρειάζεται για να ικανοποιήσει τις δικές της ανάγκες. Ακόμη και αν αυτή η παραγωγή γίνεται σε άλλο ε, χώρο από εκεί που βρίσκεται η επιχείρηση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα γραφειοκρατικό. Όποιος παράγει ενέργεια σε τόπο διαφορετικό από εκεί που το καταναλώνει, έχει πρόβλημα λογιστικό. Εάν καταφέρουμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτή την αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εφορία της Green Economy θα προχωρήσει και χωρίς να υπάρχουν πολλοί πόροι, απλά με την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Από την άλλη πλευρά τίθεται και το θέμα της μίσης, της κατανάλωσης, της ενεργειακής δηλαδή απόδοσης τόσο από τους ιδιώτες όσο και από τις δημοσίες αρχές. Όλες οι δημόσιες αρχές λοιπόν σε οποιοδήποτε διαγωνισμό δημοσιεύουν θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα και να υποχρεώνουν τον κόσμο να υλοποιεί πολιτικές μείωσης της κατανάλωσης. όλες αυτές οι απαιτήσει κατά την άποψή μας, όπως είπα και προηγουμένως, ε, όπως υπόθηκε και σε προηγούμενες ομιλίες, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν τα εδάφη, τις περιφέρειες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθημερινά χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν την ευφυΐα τους, την ταχύτητά τους στις περιοχές που βρίσκονται και να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες. Για να ολοκληρώσω θα σας παρουσιάσω δύο πτυχές. Τι έχει ήδη λάβει δηλαδή, χώρα στη δική μας ευφυή περιφέρεια. Έχουν γίνει πολλά και γίνονται πολλοί πειραματισμοί έχουν υλοποιηθεί μέσα παροχής κινήτρων για καινοτόμες επιχειρήσεις, συνεργασίες ε, για να χρησιμοποιηθούν από κοινού οι εμπειρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον τομέα της έρευνας και κυρίως στη δική μας περιφέρεια. Έχουμε μια σειρά πρωτοβουλειών για να εξάγουμε την τεχνογνωσία μας σε όλο τον κόσμο, στην Κίνα, στην Ιαπωνία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας ε, βασίζονται και σε άλλες τεχνολογίες, πολλές τεχνολογίες. Στην πράσινη τεχνολογία όπου αριστεύει η πουλια, για παράδειγμα, ε, βασίζεται και στην επεξεργασία πλάσματος, μια συγκεκριμένη τεχνολογία όπου συμβιώνει ο κόσμος της έρευνας και ο κόσμος της παραγωγής. Αυτή η τεχνολογία στην Ιταλία είναι γνωστή. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα ερευνητική στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι. Δύο έχουν εξειδικευτεί στον κόσμο, στην Ναπούλια και στη Γερμανία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πράσινης τεχνολογίας που επιτρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την αηφορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς διαφορετικής φύσης. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση στους συναδέλφους θα ήθελα να πω, επειδή χρησιμοποιήθηκαν οι διαφάνειες στα Ιταλικά, μπορείτε να βρείτε στην είσοδο την αγγλική εκδοχή. Η γραμματεία θα με ρημνήσει ώστε να προωθήσει σε όλα τα μέλη όλες τις παρουσιάσεις αυτές γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν όχι μόνο για τις σημερινή συνεδρίες αλλά γενικότερα. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας με την ομιλία τώρα της κυρία Σιμαγκουλάτα Ροντρίγκες Πινέρο Ισπανίδας βουλευτού. Έχετε τον λόγο. Δεν έχει μικρόφωνο η κυρία Φερνάντες. Συγγνώμη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να πάρω μέρος σε αυτή την ακρόαση και να μπορέσω να ακούσω τις τόσο ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις των ε, συναδέλφων που ε, μίλησαν πριν από μένα. Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο την κατάσταση και τις ανάγκες που υπάρχουν στη βιομηχανική πολιτική σε μια συγκεκριμένη περιοχή του νότου της Ισπανίας. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ τον χρόνο που μου δώσατε. Καταρχάς θα παρουσιάσω την κατάσταση της βιομηχανίας στην Ισπανία για να γνωρίζετε τα βασικά. Να συζητήσω το τι απαιτείται για την εκ νέου εκβιομηχάνηση της Ευρώπης και τοπικά τι μπορεί να είναι απαραίτητο στην Ισπανία. Καταρχάς για την κατάσταση στην Ισπανία. Να πω ότι το βάρος της, ε, το βάρος της ε, η βιομηχανία στην Ισπανία είναι γενικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην ε, Ευρώπη έχουμε ένα μέσο όρο 19,5. Ε, η βιομηχανία λοιπόν είναι λιγότερο ζυγισμένη στην ε, Ισπανία και αυτό έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, έχει περιοριστεί η δραστηριότητα, έχει να κάνει όμως βασικά με το αναπτυξιακό μοντέλο στην Ισπανία η ύφεση αυτή. Στο παρελθόν ε, βασιστήκαμε στη γεωργία και είχαμε αναπτυξιακούς ρυθμούς ε, πάνω από 10%. Στη βιομηχανία ωστόσο δεν ήταν κάτι τέτοιο δυνατόν και έτσι η πίεση μετατρέθηκε αποκλειστικά στον αγροτικό κλάδο και αυτό αποτυπώθηκε και στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Το 2011 σε ό,τι αφορά το βιομηχανικό τομέα είχαμε 20,2%. Και ύστερα, τα τελευταία χρόνια, δημορφώθηκε μια ύφεση της τάξης του 3% σε ό,τι αφορά την ε, γεωργία. Όλα αυτά φυσικά, όπως σας είπαμε, είχαν επιπτώσεις και στον τομέα της βιομηχανίας και Τώρα προσπαθούμε να δώσουμε νέα ζωή στην ε, βιομηχανία και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν, γιατί όπως ξέρετε έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ανεργία σήμερα και αυτό σε μακροπρόθεσμο επίπεδο δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Έγιναν διάφορες μελέτες λοιπόν και σε ό,τι αφορά τους ανέργους που δεν έχουν κανένα πρόσοδο και δεν έχουν καμία δυνατότητα διαφυγή για να δημορφωθεί λοιπόν μια νέα πολιτική σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία, σε ό,τι αφορά την αλλαγή τώρα του αναπτυξιακού, του παραγωγικού μοντέλου. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ισπανία εδώ και χρόνια, από το 2004, ζητά να αλλάξει το μοντέλο αυτό και ε, έχουμε υποβάλει προτάσεις για μια σχετική πολιτική που θα βασίζεται σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και βασικό, ήταν, βασικό στοιχείο ήταν και η μείωση του κόστου για τις επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, τη επιμελητία. Επίσης, ε, το θέμα ήταν η αναπτυξιακή πολιτική, η ενεργειακή πολιτική και σε όλες αυτές τις τομείς λοιπόν έπρεπε να μειωθεί η το κόστος. Το 70% του κόστους της βιομηχανίας στην Ισπανία αφορά την ενέργεια. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι... Στην Ισπανία και όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε άλλες χώρες του νότου της Ευρώπης βρισκόμαστε σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Συνειδητοποιούμε τις ανάγκες που υπάρχουν για την σωστή ανάπτυξη μιας βιομηχανικής πολιτικής. Παράλληλα με αυτές τις ανάγκες θα πρέπει να προωθήσουμε κάποιους τομείς σημαντικούς, τους οποίους πρέπει να εξυγχρονίσουμε, θα πρέπει να καταστήσουμε τους τομείς αυτούς παραγωγούς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και να μην περιοριστούμε στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα των υπηρεσιών γενικότερα, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την περίπτωση της Ισπανίας. Σας είπα λοιπόν ότι υπάρχει μια θα έλεγα σχετική αδυναμία του βιομηχανικού τομέα στην Ισπανία, αλλά παρόλα αυτά ε, υπάρχουν και κάποιες θετικές πλευρές. Ε, είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα αυτοκινήτων. Ε, έχουμε γενικά ιδιαίτερες δραστηριότητες στον τομέα των υποδομών μεταφορών, ε, έχουμε επίσης ε, ε, υψηλό επίπεδο παραγωγής εξοπλισμών για φωτοβολταϊκή ενέργεια, για αιωλική ενέργεια και έχουμε επίσης και το θέμα της γνώσης στον τομέα της διαχείρισης της, ε, των δικτύων μεταφορών και των υποδομών των μεταφορών. Δεν υπάρχει όμως μια στρατηγική πολιτική για τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι παραδοσιακοί βιομηχανικοί τομείς που έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα όπως ε, η φαντουργία, όπως η βιομηχανία τροφίμων, Αυτό δεν έχει γίνει για όλους τους τομείς βέβαια. Εμείς προωθούμε μέτρα βιομηχανικά σε οριζόντιο επίπεδο έτσι ώστε να βελτιωθούν ακόμα οι προϋποθέσεις και να ξεχωρίσουν βελτιωνόμενες όλες οι επιχειρήσεις που το αξίζουν. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο θα έλεγα γενικά. Τώρα ε, θα ήθελα να πω για την ε, βιομηχανική στρατηγική στην Ευρώπη. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι το οποίο νομίζω έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Η πολιτική αυτή δεν συνδέεται σωστά με τη μακροοικονομική πολιτική και με τις πολιτικές λιτότητας και εξυγίανσης δημοσιονομικής. Είναι δύσκολο να προχωρήσει κανείς σε μέτρα στα πλαίσια της πολιτικής ε, εκβιομηχάνησης όταν από την άλλη η πολιτική λιτότητα οδηγεί στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στη συρρήκνωση κάποιων τμήματων της βιομηχανικής δραστηριότητας. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα ελλείμματα. Εμείς ε, είμαστε υπέρ των επενδύσεων σε κάποιες παραγωγικές δραστηριότητες, θέλουμε επενδύσεις και στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, γιατί αυτές οι δύο πολιτικές είναι απαραίτητες για να γίνουμε ακριβώς πιο ανταγωνιστικοί και να βγούμε από την ύφεση. Δεν μπορούμε να περάσουμε επίσης σε μία εκ νέου εκβιομηχάνηση των περιοχών μας σε δύο ταχύτητες, με δύο ταχύτητες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε. Δηλαδή ε, χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλή αμοιβή, ε, χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο σε κάποιες περιοχές και υψηλές τιμές, υψηλά επίπεδα αμοιβών κτλ. σε άλλες χώρες. Υπάρχουν χώρες βέβαια οι οποίες έχουν ε, λιγότερους ε, ανέργους, από την άλλη έχουν πάρα πολύ χαμηλούς ε, μισθούς. Εμείς αντίθετα θα πρέπει νομίζω να αλλάξουμε τις συνθήκες αυτές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το πετύχουμε αυτό είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σωστά στον τομέα της κατάρτισης της επαγγελματικής από τη μία και της κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών από την άλλη. Ε, το κόστος στην Ισπανία οι προσπάθειες αυτές είναι, για τις προσπάθειες αυτές είναι πάρα πολύ υψηλό είναι το κόστος πολύ πιο υψηλό, υψηλό το κόστος σαν παράδειγμα δανειοδότησης ορισμένων δραστηριοτήτων και με τόσο υψηλό χρηματοδοτικό και ε, επενδυτικό κόστος ε, για τις επιχειρήσεις μας ε, τα πράγματα δεν είναι καλά και οδηγούν σε πολυδιάσπαση των αγορών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε λοιπόν και σε εθνικό επίπεδο να θέσουμε ακριβώς αυτή την πορεία προς την εκ νέου ε, και βιομηχάνηση της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς εμείς σαν πολιτικό κόμμα ασκούμε κριτική στις ε, ρυθμίσεις και στα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση της χώρας ε, αποδυναμώνει τις πολιτικές τις οποίες θέλουμε ακριβώς να προωθήσουμε. Δεν μπορεί να συνεχίσει η κατάσταση. Εμείς είμαστε αντίθετοι με την πολιτική αυτή. Θέλουμε να προωθήσουμε μια μεταρρύθμιση φορολογική η οποία θα δώσει τα μέσα για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αυτό θα πρέπει να υπάρξει θα έλεγα μια προσπάθεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην υπάρχουν εντελώς διαφορετικές φορολογικές βάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έτσι ώστε να υπάρξει ένα ισότιμο πεδίο ανάπτυξης για τη βιομηχανία. Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε και την διεθνοποίηση των ε, βιομηχανικών επιχειρήσεων για περισσότερες ε, εξαγωγές. Πρέπει να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις αυτές, οι τομείς αυτοί έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα κάποιες επιχειρήσεις ε, να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες και να μην υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ τους. Εδώ να σημειώσω επίσης ε, και το θέμα της ευθύνης των επιχειρήσεων. Δηλαδή πώς μπορούν να πάρουν μέτρα οι επιχειρήσεις οι ίδιες έτσι ώστε να εμπλέξουν στην καθημερινή λειτουργία τους τους εργαζομένους τους και να εκπαιδεύσουν και να καταρτήσουν σωστά τους εργαζομένους. Τίθεται το θέμα της ευθύνης δηλαδή των επιχειρήσεων και του πλαισίου του νομικού σε κάθε χώρα. Έτσι θα γίνουμε παραγωγικοί, έτσι θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Τελευταίος ομιλητής σε αυτό το πάνελ είναι ο κύριος Γιάνσεν. Ε, thank you, thank you, Chair. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε την ΕΤΟΚ, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων, να ε, σας παρουσιάσει τις απόψεις της για το θέμα αυτό. Από πλευράς ΕΤΟΚ θα πρέπει να σας πούμε ότι ε, μας απασχολεί το θέμα αυτό Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω επενθυμίζοντας κάποια βασικά γεγονότα. Καταρχάς ότι η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία από την περίοδο από το 1998 μέχρι το 2009 έχει χάσει 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 17% περίπου της βιομηχανικής απασχόλησης που έχει χαθεί σε περίοδο δεκαετών. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε όχι μόνο αυτά τα στοιχεία, αλλά και άλλη μία ε, τάση που προδιαγράφεται εκ παραλλήλου, μία τάση της βιομηχανίας να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, εδώ δίνω το παράδειγμα, γιατί είναι και το κατεξοχήν παράδειγμα της επιτυχίας, το παράδειγμα της Γερμανίας. Η Γερμανία το 1998 είχε 17,6% του συνολικού μεριδίου, αν θέλετε, των βιομηχανικών θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη, 35 εκατομμύρια περίπου. Τώρα όμως έχει το 19,3%. Πρόκειται λοιπόν για μια ένδειξη ε, επιτυχίας η οποία αυξάνεται σε σημασία κοιτώντας και τον υποτομέα των ε, μηχανημάτων που είναι πολύ σημαντικός τον υποτομέα λοιπόν εξοπλισμού και μηχανημάτων που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτός είναι σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ σημαντικός σε ό,τι αφορά τη Γερμανία. Κοιτώντας λοιπόν τα επίπεδα του 1998, τότε η Γερμανία είχε 26% του ποσοστού αυτού. Το 2009 το ποσοστό αυτό είχε ανέλθει από 26% στο 33%. Άρα το 1 τρίτο των θέσεων απασχόληση σε ό,τι αφορά τον υποκλάδο αυτό εξοπλισμού και μηχανημάτων είναι σε συγκεκριμένες περιφέρειες της Γερμανίας. Αυτό νομίζω ότι εξηγεί γενικότερα την πολύ καλύτερη γερμανική απόδοση από ό,τι άλλες χώρες της Ευρώπης. Κοιτώντας λοιπόν τώρα τα ποσοστά απασχόλησης και κοιτώντας, περνώντας από τα ποσοστά απασχόλησης στα ποσοστά προστιθέμενης αξίας, η εικόνα είναι παρόμοια. Βλέπουμε λοιπόν την προστιθέμενη αξία της ε, ε, γερμανικής μεταποιητικής βιομηχανίας ως ποσοστό του ΑΕΠ και την τάση που διαγράφεται τα τελευταία χρόνια και με την κρίση, την ανάκαμψη μετά την κρίση του 2009, η Γερμανία βρίσκεται στο στο έχει πετύχει το στόχο αυτό του 20% του, μετα, της μεταπητικής βιομηχανίας που συζητάμε εδώ. Κοιτάτε, και βλέπουμε την άλλη γραμμή, η τάση που διαγράφεται στην Ευρώπη είναι πτωτική και κοιτώντας περαιτέρω λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις χώρες της Ευρωζώνης, τις χώρες του Νότου ιδιαίτερως, βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση σε ό,τι αφορά τη μεταπητική βιομηχανία, ιδιαίτερα στην Ισπανία, στη Γαλλία. Επίσης είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και χαμηλό το ποσοστό, περίπου 12% σε ό,τι αφορά το ποσοστό συμμετοχή στο ΑΕΠ και σε χώρε όπω η Ελλάδα είναι και κάτω από το 10% ακόμα το ποσοστό αυτό, 8% σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή δηλαδή τη μεταπητική βιομηχανία. Ωστόσο στην Ιταλία είναι αυξητική η τάση Παρ' όλα αυτά όμως το επίπεδο εξακολουθεί να είναι γύρω στο 16% που είναι, σημαίνει δηλαδή ότι είναι δεύτερη στη σειρά μετά τη Γερμανία. κοιτώντα λοιπόν τη Νότια Ευρώπη οι α, διαφορές είναι πολύ μεγαλύτερες. Η Ισπανία δεν είναι ίδια με την Ιταλία, ούτε η Ισπανία είναι ίδια με την Πορτογαλία και δυστυχώς η Ελλάδα είναι και ακόμα πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Και γιατί λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρξει, να διατηρηθεί σε ένα κράτος μέλος, σε όλα τα κράτη-μέλη αυτή η βιομηχανική, η μεταπητική βάση. Για δύο λόγους. Γιατί η ισχυρή βιομηχανική βάση ε, συνεπάγεται κατά κανόνα υψηλότερη ε, προστιθέμενη αξία, θέσεις απασχόλησης, υψηλότερους μισθούς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν μας απασχολεί η κοινωνικο-οικονομική συνοχή στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε αντίστοιχη ισχυρή βιομηχανική βάση σε πολλές περιφέρειες και χώρες στην Ευρώπη. Ιδάλλως θα αυξάνονται οι ανισότητες στο εσωτερικό της Ευρώπης. Ένας άλλος λόγος έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή κρίση, γιατί μια ισχυρή βιομηχανική βάση δίνει σε μια χώρα τις εξαγωγές που χρειάζεται για να πληρώσει τις εξαγωγές της. Χωρίς αυτή τη βάση και με τα τρέχοντα ελλείμματα ισολογισμών κατάσταση διαμορφώνεται προβληματική, γιατί ουσιαστικά χρειάζεται αύξηση του δημόσιου χρέους. Άρα, με άλλα λόγια, με τα τεράστια ελλείμματα της τελευταίας δεκαετίας σχηματίστηκαν τεράστια χρέη, δημόσια χρέη, τεράστιες φούσκες χρηματοπιστωτικές και αυτό αποτελεί την πηγή της ευρωπαϊκής χρήσης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν θέλουμε να σώσουμε το ευρώ, αν θέλουμε να λύσουμε την κρίση, θα πρέπει να υπάρξει τέτοια βιομηχανική βάση και στο νότο της Ευρώπης. Δεν θα ήταν σωστό στην παρούσα φάση να πούμε ότι δεν υπάρχει καθόλου στρατηγική επαναβιομηχανοποίηση στο νότο της Ευρώπης. Αντιθέτως, κοιτάζοντα τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ τα προγράμματα τη Τρόικα, διαπιστώνουμε ότι ένα από του κρυφού ίσω στόχου είναι πράγματι η εκ νέου βιομηχανοποίηση του Νότου με την πολιτική ε, ευέλικτης διαμόρφωσης όλων των τομέων του τομέα απασχόλησης, ε, των επιδομάτων ανεργίας, ε, των κοινωνικών επιδομάτων. Όλα αντιμορφώνονται με πιο ευέλικτο τρόπο και σκοπός είναι να καταστούν ανταγωνιστικά ως πρωτοκόστος αυτά τα κράτη-μέλη με απόλυτο αλλά και σχετικό τρόπο προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις. Όπως είδαμε υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με αυτό. Αυτό έχει να κάνει και με αμφιβολίες σε μακροπρόθεσμο ε, επίπεδο, γιατί πρόκειται για μια στρατηγική γενικής πτώχευσης, αν θέλετε. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να διατηρηθεί μια ισχυρή βιομηχανική βάση, ε, μειώνοντας το βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού, κλείνοντας τα σχολεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε μακροπρόθεσμα ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, ε, ένα άλλο φαινόμενο είναι η μαζική μετανάστευση, ιδιαίτερος των ε, εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης και αυτό φυσικά καταστρέφει τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ισχυρής βιομηχανικής βάσης. Τι θα πρέπει λοιπόν να αποτελεί την εναλλακτική λύση. Μία στρατηγική ευελιξία, στην οποία και προασπίζουμε μια στρατηγική προσπίζουμε μια στρατηγικη επενδυσεων που αναπτύσσει τα προϊόντα εκείνα, τις ε, δραστηριότητες, τους τομείς εκείνους, βάσει των οποίων τα κράτη-μέλη του Νότου μπορούμε να πούμε ότι έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Τι έχουμε υπόψη μας, η παραγωγή, για παράδειγμα, βιώσιμης ενέργειας, όπου ο Νότος έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η φιλοσοφία λοιπόν που κρύβεται πίσω από τη στρατηγική αυτή είναι η εξή. Επενδύοντα στου τομεί αυτού, αναπτύσσοντα τι υπηρεσίε και τα προϊόντα αυτά, δίνουμε στι χώρε αυτέ μία βάση εξαγωγή. Και έτσι δημιουργούν έσοδα, αποπληρώνουν τα χρέη τους στις βελγικές, γερμανικές, γαλλικές ε, τράπεζες και έτσι πέρα από αυτό τα κράτη-μέλη αυτά έχουν δραστηριότητα, διατηρούν θέσεις εργασίας. Είναι πολύ διαφορετική λοιπόν η στρατηγική αυτή που εστιάζεται στη μείωση του βιωτικού επίπεδου, στην ε, περιορισμό των θέσεων απασχόλησης. Ποιες δραστηριότητες και ποια προγράμματα έχουμε υπόψη μας. Τέσσερα βασικά μπορούμε να τα πείσουμε. Βλέπετε στη διαφάνεια ότι ένα βασικό στόχος είναι η οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτροδότησης με τις βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Νότου. Αυτό θα ήταν ε, πολύ καλό για τις χώρες αυτές. Ένα δεύτερο είναι ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα για την ε, δημιουργία δικτύων μεταφοράς υψηλής απόδοσης αλλά και ε, ευρυζωνικών δικτύων. Ένας τρίτος τομέας είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για ε, επενδυτικέ επιδοτήσεις ή δάνεια χαμηλών επιτοκίων σε εταιρείε οι οποίες μπορούν να δαπανίσουν με τη σειρά του σε ενεργειακές ε, χρήσεις υψηλής αποδοτικότητας και έχουμε το σχετικό ίδρυμα στο Βερολίνο που υπολογίζει 300 δισεκατομμύρια δυναμικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά δηλαδή, την βελτίωση της αποδοτικότητας των δικτύων ε, ηλεκτροδότησης και παροχής ενέργειας. Τέταρτο στομέας, ένα πρόγραμμα μικροπιστώσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάρα πολύ σημαντικό γιατί στις ε, τρέχουσες στάσεις που διαμορφώνονται στην Ευρώπη, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοια προγράμματα για το νότο της Ευρώπης, για τις επιχειρηματικές δομές στο νότο της Ευρώπης. Στην τελευταία διαβάνεια, πρόεδρε, που έχω φέρει, επιμένουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και θα πρέπει η χρηματοδότηση επίσης να έρχεται από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γιατί, γιατί τα κράτη του Νότου είναι τα πιο ευάλωτα από οικονομικής άποψης. Δεν μπορούν να δώσουν τους πόρους αυτούς από μόνα τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια, ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα που θα κατευθύνονται όλος ιδιαίτερος προς, τα, προς τις αδύναμες αυτές τις περιφέρειες που χρειάζονται την ενίσχυση. Όπως βλέπετε έχουμε βάλει και ένα συγκεκριμένο ποσοστό, έχουμε ορίσει ένα ποσοστό το οποίο ασφαλώς μπορεί να προσαρμοστεί. Εμείς θεωρούμε ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να κυμαίνεται στο 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ σε ό,τι αφορά δηλαδή τα κονδύλια που θα δαπανηθούν προς τις στρατηγικές αυτές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς και αυτή η παρουσίαση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Σε αυτό το παράλληλο έχουν γίνει πολλές αιτήσει για ομιλητές. Ξεκινάμε από τον κύριο Πιτικόφερ, τον κύριο Σιγητή. Δύο λεπτά θα έλεγα για όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω τρεις ερωτήσεις για τον τελευταίο ομιλητή της TUC. Ξεκινώντας από το τελευταίο σημείο που αναφέρατε Ευρωπαϊκή επενδυτική χρηματοδότηση 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ δεν με πείθει έτσι εύκολα δεδομένου ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχει κίνδυνος να πέσει κάτω από το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Θα μπορούσατε λοιπόν ενδεχομένως ε, να μας βρείτε μια μαγική λύση για αυτό το πρόβλημα ή μήπως θα μπορούσε το ETUC να υπερασπιστεί έναν διαφορετικό προγραμματισμό για το πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν έχω εγώ ακούσει πρόσφατα. Δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά τη δική σας στρατηγική σε σχέση με την ενέργεια και την αποδοτικότητα των πόρων, Συμφωνώ απόλυτα, αλλά περιορίσατε τις προτάσεις σας σε επενδυτικές χορηγίες και δάνεια χαμηλών επιτοκίων. Μπορείτε να φανταστείτε και κάποια άλλα εργαλεία σε αυτή την εργαλειοθήκη, όπως αλλαγή των κανονιστικών ρυθμίσεων των αγορών για την πρόθεση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Τι από αυτά θα ήσασταν διατεθειμένοι να υιοθετήσετε. Τρίτον, δεν ε, επικεντρωθήκατε ιδιαίτερα στο ζήτημα των δεξιοτήτων. Πολλές συζητήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με τα πλεονεκτήματα της διπλής επαγγελματικής, των διπλών συστηματών επαγγελματικής κατάρτισης που ορισμένες χώρες ε, εφαρμόζουν εδώ και καιρό και που άλλες χώρες τώρα τολμούν να υιοθετήσουν. Πώς το βλέπετε αυτό στην ETUC, θα μας βοηθήσετε να προωθήσουμε αυτά τα διπλά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η συνάδελφος Αντρές Μπαράγια, σκιώδης των σοσιαλιστών για την έκθεση αυτή για την εκβιομηχάνηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας και τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πράγματι περιμένουμε πολλά από τις καινοτομίες και τίθεται φυσικά και το θέμα της ε, ενέργειας. Εκεί έχουμε κάποια προβλήματα, δεν έχουμε καθορίσει ακριβώς την πορεία προς τη λύση που είναι ένα ευρωπαϊκό και μια ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας. Τίθεται φυσικά κυρίως και το πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα για τις χώρες του Νότου, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και πάρα πολλοί έχουν αρχίσει να μιλάνε για τον γερμανικό κίνδυνο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι θέμα αξιολόγησης. Ε, τώρα σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής μας ο κύριος Μποτικόφερ, που λέει ότι ίσως να χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση για τις χώρες του Νότου. Εγώ εδώ νομίζω ότι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υπάρξει μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση, διότι αυτό σημαίνει ε, μια ρήξη στην Ευρώπη, μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων την οποία δεν μπορούμε να αποδεχθούμε και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο δημοκρατίας. Αυτό που απαιτείται είναι να υπάρξει μια διαφοροποιούμενη μορφή χρηματοδότηση. Είναι σαφές ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές έχουν έχει τεθεί το θέμα της μείωσης ε, του ΑΕΠ. Ε, δεν εφαρμόζονται οι αντιλήψεις ε, σχετικά με την αλληλεγγύη, την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία προτείνει το Συμβούλιο. Τίθεται όμως το θέμα της συγχρηματοδότησης. Πολλές φορές οι χώρες δεν μπορούν να δίνουν το 50% για κάποια προγράμματα και κάποια προγράμματα απλά δεν προχωρούν. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με περιοριστικούς όρους, θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει και λύση για την σωστά προσανατολισμένη χρηματοδότηση, στοχευμένη χρηματοδότηση, όχι γενικά τη χρηματοδότηση χωρών. Έτσι θα ωφεληθεί η βιομηχανική πολιτική, η οποία είναι ουσιαστική για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση. Αλλά θα πρέπει η χρηματοδότηση αυτή, όπως είπα, να είναι σωστά προσανατολισμένη. Λάγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Μαντουέλε που δεν, θα μπορέσει να παραστεί σήμερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε θέματα ε, ε, ε των βιομηχανιών της ε, Νότιας Ευρώπης ποιοι είναι οι παράγοντες που παίζουν ε, ρόλο πέρα από το μισθολογικό κόστος. Είπε η συνάδελφος από την Ισπανία ότι η επικέντρωση και μόνο στο μισθό και στο μη μισθολογικό κόστος δεν μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, αλλά ουσιαστικά συνεχίζει το φαύλο κύκλο προς τα κάτω. Θα πρέπει λοιπόν να εκτιμήσουμε και τους άλλους παράγοντες που έχουν σημασία. Το θέμα που αντιμετωπίζει και η Γερμανία και η Σουηδία το θέμα της καινοτομία, το θέμα του κοινωνικού διαλόγου και στη Γερμανία και στην ε, Σουηδία ε, μιλάμε για χώρες με παράδοση στον κοινωνικό διάλογο και σε ό,τι αφορά τον ορισμό των κοινών στρατηγικών για την βιομηχανία. Άρα λοιπόν, ιδιαιτέρως από πλευρά της Ισπανίας, αλλά και από την πλευρά της ΕΤΟΚ, θα ήθελα να ακούσω ποιοι πιστεύουν ότι είναι οι άλλοι παράγοντες, πέρα από το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος, που τελικά επηρεάζουν και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, πέρα από την καινοτομία δηλαδή, πέρα από το θέμα του κοινωνικού διαλόγου και το θέμα των ικανοτήτων. Βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο μόνο 29% των εργαζομένων έχουν πρόσβαση σε τέτοια εκπαίδευση και σε ό,τι αφορά την εκ νέου κατάρτιση, μόνο 7% είναι το ποσοστό αυτό. μήπω και αυτό επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα. Αυτά θα ήθελα να ακούσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να αναφερθώ στην παρουσίαση του συναδέλφου κυρίου Μπράτα και να επισημάνω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, θα μπορούσαν να συνδεθούν με το πρόβλημα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή όλα τα θέματα που αφορούν ε, ειδικότερα αφενός ε, τη χρήση των ε, δασικών και γεωργικών απορριμμάτων, τη βιομάζα και τη διατήρηση των υδατινών πόρων και τα μικρά υδραυλικά συστήματα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να επισημανθούν. Δεύτερον, όσον αφορά την παρουσίαση του κύριου Γιάνσεν, την βρίσκω εξαιρετικά σημαντική. Θεωρώ ότι το 2% είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην σε μια λύση από αυτή την ε, στασιμότητα, για να μην πω οπισθοχώρηση. Σαφώς ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι εκείνη που άμεσα ή έμεσα θα δημιουργήσει τέτοια κονδύλια, θα τα κάνει διαθέσιμα, διότι διαφορετικά δεν πιστεύω ότι η Ιταλία του Νότου η Νότια Ευρώπη γενικότερα θα μπορέσει να ανακάμψει σε θέματα ανταγωνιστικότητας ακόμη και αν εμείς μισθοί παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Για να απαντήσω δηλαδή στο συνάδελφο κ. Μπουτικόφερ, ελπίζω ότι οι ευρωεκλογέ ε, θα μας δώσουν κάποια ελπίδα ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε Eurobonds ή Project Bonds ε, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να αφιερωθούν σε αυτό το στόχο. Συνάδελφος Τράουτμαν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τις επενδύσεις. Πολλοί από εσάς ε, αναφέρατε την προβληματική της ενέργειας και των δικτύων. Κοιτώντας σήμερα το ζήτημα των δικτύων, εγώ διαπιστώνω ότι έχουμε ανεπαρκείς επενδύσεις, ανεπαρκή χρηματοδότηση και στάση παράδοξη μεταξύ των πολιτικών στην Ευρώπη. Η συζήτηση που είχα πρόσφατα με την Επενδυτική Τράπεζα για τα δίκτυα ψηφιακής τεχνολογίας δείχνει ότι το κόστος της πίστος σε αυτούς τους τομείς είναι υψηλότερο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρεί ότι είναι πιο ρηψοκίνδυνε αυτέ οι επενδύσει από ό,τι στι μεταφορέ ή στην ενέργεια. Και εγώ ρώτησα, μπορούμε να βρούμε κάποιον τρόπο να, να ευνοήσουμε αυτού του είδου επενδύσει. Είναι σαφή η απάντηση. Χρειάζονται δημόσιε εγγυήσει. Αυτό που είναι σαφέ λοιπόν ότι για να, βγούμε, να βρούμε μια λύση πρέπει να φέρουμε τη συζήτηση αυτή με το τέλο. Δεν μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική και μέσα που δεν λειτουργούν. Αυτή είναι μια διαπίστωση αναμφίβολη. Οι επενδυτικές επιχειρήσεις έρχονται εκεί όπου υπάρχουν χαμηλές τιμές ε, κατανάλωσης ενέργειας, ε, όπου υπάρχουν συστήματα παροχής ενέργειας, ειδικότερα στο βιομηχανικό τομέα, ειδικότερα για κάποιες βιομηχανίες που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και φυσικά χρειάζονται συνδέσεις με τα δίκτυα πολύ υψηλής ταχύτητας. Γνωρίζουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις και εγώ θεωρώ ότι σε σχέση με τον Νότο Κάποια στιγμή με τον Ζακ Ντερόλ δημιουργήσαμε τα διαρθρωτικά ταμεία ώστε να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε να... την ανάπτυξη και να προσφέρουμε έναν επιταχυντή. Και εγώ προτείνω και θα ήθελα να μου απαντήσουν τα μέλη του πάνελ εδώ γιατί πρόκειται για μια δύσκολη μάχη. Πρόκειται για μια πρόταση που έχει ήδη γίνει αλλά που δεν έχει γίνει δεκτή από το Συμβούλιο ούτε απολύτως από το δικό μας Κοινοβούλιο. Εγώ προτείνω να έχουμε αποτελεσματικά προγράμματα σε αυτούς τους τρεις τομείς δικτύων, μεταφορές, ενέργεια, επικοινωνία και πληροφορική, όπως προτάθηκε αλλά με περισσότερα μέσα και προτείνω για το ρόλο που θα διαδραματίσουν σε αυτές τις επενδύσεις τα κράτη-μέλη να αφαιρέσουμε από τον υπολογισμό του δημοσίου χρέους τους τις επενδύσεις σε αυτού του είδους τα δίκτυα. Εγώ πιστεύω ότι κάτι είναι απολύτως αναγκαίο. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει δημόσια εγγύηση για ιδιωτικές επενδύσεις. Μπορείτε να δείτε σήμερα το πρόγραμμά μας είναι αστείο. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τις διασυνδέσεις ε, στον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνίων δεν αξίζει καν να το συζητάμε. Δεν αρκεί ούτε για μια μικρή χώρα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι σοβαρό. Αναφέρθηκε για τους νέους. Το πρόβλημα των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των ανθρωπίνων πόρων. Εγώ ανα... αμφιβάλλω για αυτή όπου λέμε ότι πρέπει να ευνοήσουμε την κινητικότητα των νέων. Πολύ καλά το κάναμε με το Εράσμους, αλλά πιστεύω ότι εδώ οργανώνουμε αποκέντρωση των ανθρωπινών πόρων και απόλυτη ανταγωνιστικότητα σήμερα, διότι ένας νέος που δεν αξιοποιεί τις ικανότητες του για τρία-τέσσερα χρόνια θα τις χάσει και θα γίνει πολύ λιγότερο αξιόπιστο στον αγορά εργασία. Υπάρχουν πολλέ δυνατέ λύσει φυσικά. Θα πρέπει να μελετήσουμε αυτή την πρωτοβουλία για του νέου. Αλλά πιστεύω ότι μια πρόταση που είχε γίνει στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων το να συνδυαστούν παγκόσμιοι πόροι έρευνα και καινοτομία ε, με πλατφόρμες στις χώρες του Νότου, αυτή είναι μια λύση που θα μπορούσε να υλοποιηθεί πολύ γρήγορα. Υπάρχουν ήδη τα σχετικά προγράμματα και πιστεύω ότι θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βρούμε τις σχετικές λύσεις ώστε να υπάρξει ανάκαμψη των επιχειρήσεων. Και το τρίτο που ήθελα να πω, πιστεύω τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι έγινε με αυτό το 3% του ΑΕΠ που θα είχαμε για την έρευνα και την καινοτομία. Δεν το συζητάμε πια σήμερα το, στο οποίο θα βασιζόταν η ανάπτυξη των χωρών μας. Δεν φτάσαμε ποτέ αυτό το 3% γιατί δεν είχαμε τα μέσα. Και εγώ αυτό που έχω να σας πω επ' αυτού είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ότι οι μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις όταν συγκεντρώνονται είναι ικανές να επιτύχουν ανάκαμψη. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, η κεφαλαιοποίηση και η πρόσβαση σε πιστώσεις. Εσείς το είπατε και εγώ να ρωτιέμαι. Έχουμε την καινοτομία, τα νέα προϊόντα, τον νέο τρόπο διοργάνωσης των βιομηχανικών διαδικασιών, αλλά υπάρχει και η ανάκαμψη η δυνατότητα μιας περιοχής χαρακτηρίζεται από την επιτυχία των επιχειρήσεων της περιοχής. Και τι γίνεται όταν αποσύρονται οι διεθνείς επενδύσεις. Πιστεύω ότι οι στρατικές μας είναι ανεπαρκείς σε αυτό. Επίσης πιστεύω, τέταρτον, ότι στους δημόσιους διαγωνισμούς θα μπορούσαμε να εισάγουμε ρήτρε που να ευνοούν την, εισαγωγή, την ένταξη των νέων, ώστε οι επιχειρήσεις που κερδίζουν δημόσιους διαγωνισμούς να μπορούν να προσλαμβάνουν νέους, να τους δίνουν δουλειά. Δεν αρκεί για να λύσουμε το πρόβλημα της ενέργειας των νέων, αλλά θα μπορέσει να βοηθήσει και θα μπορούσε επίσης να αποτελεί και μια ευρωπαϊκή πολιτική ευνοϊκή που θα συμβάλλει στις όλες κοινέ προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο συναδελφός Ευχαριστώ Πρόεδρε κάποια επιπλέον στοιχεία. Βρισκόμαστε στο δεύτερο πάνελ, εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι απαιτείται μια εκ νέου ε, βιομηχάνηση του Νότου, διότι το πρόβλημα της βιομηχανίας είναι σφαιρικό και βρισκόμαστε σε ανταγωνισμό με άλλες περιοχές του κόσμου. Για τον κύριο Μπράτα, πράγματι θέσατε το θέμα της γραφειοκρατίας και των νομικών περιορισμών. Αυτή η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και σε εθνικό επίπεδο η γραφειοκρατία και πολλές φορές και σε περιφερειακό είναι απαράδεκτη. Ας αναπνεύσουν οι επιχειρήσεις μας. Οι επιχειρήσεις μας τι θέλουν, θέλουν σταθερότητα. Κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές και αλλάζουν υπουργοί, αλλάζουν και οι κανόνες. Ας σταματήσουμε λοιπόν αυτή τη διακανονιστική τρέλα. Κυρία Ροντρίγκες, Είπατε ότι δεν θα πρέπει να συνεχίσει η, Ισπανία και η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εμείς στη Γαλλία έχουμε πραγματικά 300 ε, πτωχεύσεις την ημέρα. Αν έχετε κάποια μαγική συνταγή, ε, κοιτάξτε να μας τη δώσετε. Εσείς μιλήσατε για τη λιτότητα και τα λοιπά. Πράγματι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη βασισμένη πάνω στα δημόσια έσοδα. Αυτό δεν είναι λιτότητα έτσι όπως την προέβλεπε ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Απαιτείται δημοσιονομική πειθαρχία ως προς το σοβαρό της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της δημόσιας δαπάνης. Αυτό είναι το νόημα της κρίσης. Και τώρα μια ερώτηση προς τον κύριο Γιάνσεν. Χαίρομαι για την παρουσία του οι στατιστικές της Ένωσης είναι γνωστές. 8% του παγκόσμιου πληθυσμού, 23% του πλούτου στον κόσμο και 50% της δημόσιας δαπάνης. Αυτό είναι το θέμα. Τι θα κάνουμε λοιπόν με τον κόσμο έτσι όπως είναι σήμερα. Θα ήθελα να μας εξηγήσει το γιατί δεν έχει υπάρξει περαιτέρω ε, κοινωνική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παλαιά κομμουνιστικές χώρες είναι μέλη της Ένωσης εδώ και 9 χρόνια, όχι εδώ και 9 μέρες, και όμως έχουμε μισθούς στις χώρες αυτές 100, 200 και 300 ευρώ. Στην Πορτογαλία 400 ευρώ, η σύντροφός μου είναι Πορτογαλίδα. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, να δημιουργήσουμε την ευρωπαϊκή ελπίδα όταν είμαστε ανίκανοι και σε επίπεδο εργοδοσίας και σε επίπεδο συνδικάτων και σε επίπεδο πολιτικής σε 10 χρόνια να προχωρήσουμε σε ένα ελάχιστο ποσοστό κοινωνικής σύγκλησης. Πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Και πάντα σε όλο τον κόσμο, στις σχολές, στις εμπορικές, τι λέμε. Ότι θα πρέπει οι κανόνες οι κοινωνικοί να οδηγούν στη σύγκληση. Εμείς δεν το πετύχαμε αυτό. Αυτό που είπατε εσείς για τον κοινωνικό διάλογο είναι πάρα πολύ σωστό. Θα πρέπει να δούμε σε επίπεδο κοινοτικού διαλόγου τι πηγαίνει καλά για να προχωρήσουμε μέσω αυτού. Ένα επιπλέον θέμα προς τα πάνελ. Δεν αναφερθήκαμε στις εμπορικές πολιτικές. Η φαντουργία μας στη Γαλλία καταστράφηκε επί τη βάση των εξαιτίας μάλλον των εμπορικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Μήπως είμαστε ανόητοι τελικά σε σχέση με τις πολιτικές αυτές. Όταν ο Πασκάλα μη τελειώσει ε, την περίοδο εντολής του στον Ποένα μας πει τι έχει γίνει, τι συμβαίνει. Εμείς πιστεύαμε στην πολυμέρεια και από την άλλη έχουμε εκατοντάδες εμπορικές συμφωνίες και εμείς επίσης έχουμε υπογράψει πάρα πολλές διμερείς εμπορικές συμφωνίες χωρίς αποτέλεσμα. Μήπως θα έπρεπε να προστατευθούμε καλύτερα σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τους κανόνες υγιεινής, σε σχέση με τους κανόνες που επιβάλλουμε εμείς τους παραγωγούς μας και σε σχέση με τον ανταγωνισμό όλων αυτών των υπήρων που πραγματικά εδώ και 10-15 χρόνια βλέπουμε να εκρήγνεται. Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κτλ. Μήπως η εμπορική πολιτική μας θα έπρεπε να καταστεί ένα μέσο αποτελεσματικότερο φροντίδας των δικών μας παραγωγών και όχι τόσο των καταναλωτών. Έχει το λόγο και ο Λάγκες. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν μιλάμε για την εκνεύγιο μηχανοποίηση του νότου της Ευρώπης θα πρέπει να αναλύσουμε και τις ε, παράλληλες ε, παρόμοιες διαδικασίες. Θεωρώ ότι ίσως ο καλύτερος παραλληλισμός είναι η οικονομική και κοινωνική ε, παρακμή της Δανίας το 19ο αιώνα μετά την απώλεια της Νορβηγίας, του στόλου, τη χρεοκοπία του κράτους η Δανία ήταν σε πολύ δύσκολη θέση Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Δανίας είναι ότι σήμερα τουλάχιστον έχει δύο ευφυείς άνδρες στην πολιτική ε, ζωή, τον βασιλιά και τον ε, αρχιεπίσκοπο Γκρούντβικ. Uh, uh, Αντιλήφθησαν ότι στην Ευρώπη υπήρχε ε, η τάση της αστικοποίησης, η ανάπτυξη των πόλεων. Αυτή λοιπόν προαπαιτούσε την ύπαρξη τροφίμων. Αυτό ήταν μια μοναδική διαπίστωση για την Δανία, γιατί δεν είχαν πρωτεσίλες, δεν είχαν άλλους πόρους πέρα από την παραγωγή τροφίμων. Σήμερα λοιπόν ε, έχουν συνδυάσει πλέον τα μικρά κεφάλαια σε συνεταιρισμούς και έχουν διαμορφώσει έτσι μεγάλη κεφάλαια. Έχουν ιδρύσει ένα σύστημα κατάρτισης γεωργικής εκπαίδευσης και έχουν σήμερα εταιρείες που αρχικά ξεκίνησαν από συνεταιρισμούς και έχουν ξεκινήσει εξαγωγή τροφίμων στην υπόλοιπη Ευρώπη προκειμένου να παρέχουν τρόφιμα στις, αναπτυσσόμενες, στις ε, όλο ένα και αυξανόμενε ε, σε, μέγεθο μέγεθος πόλης της Ευρώπης. Το πρόβλημα στην Νότια Ευρώπη είναι η χαμηλή ποιότητα σε ό,τι αφορά το εργατικό δυναμικό. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία, σε κάποια τμήματα της Ιταλίας και της Πορτογαλίας αυτό είναι σαφές. Και λοιπόν αυτή, αυτό το επίπεδο των ε, προσόντων του εργατικού δυναμικού είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της ε, Νότιας Ευρώπης. Ρωτώ λοιπόν να μας πει ο κύριος Γιάνσεν κάποιες ιδέες ενδεχομένως για τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν για να αυξήσουν το επίπεδο των προσόντων του εργατικού δυναμικού στα τμήματα αυτά της Ευρώπης ως ένα βασικό παράγοντα οικονομικής ανάκαμψης. Μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για κάποια μέτρα που έχουν να κάνουν με βιομηχανικά προγράμματα. Θεωρώ όμως ότι το εργατικό δυναμικό είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε ένα λεπτό τώρα δίνω στους ομιλητές για να μπορέσουν να απαντήσουν. Σας παρακαλώ να μην πάρουμε περισσότερα από τρία λεπτά ώστε να μην... Να, έχουμε περιθώριο και για τους υπόλοιπους. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομος στις απαντήσεις, μου λέει ο κύριος Μπράτο. Υπάρχουν κάποια κοινά κεφάλαια. Το πρώτο αφορά τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις στη δίκτυα είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη του τομέα αυτού. Αυτό είναι σίγουρο. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν εφαρμογής πόρων, χρήσης πόρων είναι για την ανάπτυξη των δικτύων. Πόσο μάλλον στα δίκτυα, στα κέντρα κατανάλωσης ενέργειας. Η βιωσιμότητα αυτού του τομέα δεν βασίζεται σε επιχορηγήσεις χαμένες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν μόνο κονδύλια, ζητούν διευκόλυνση της φορολόγησης και σίγουρους και απλούς κανόνες σε όλα τα κράτη. Μίλησε ο συνάδελφο για την γραφειοκρατία. Στην Ιταλία πράγματι χρειάζονται 30 άδειε για μια μικρή επένδυση. Αυτό η αρχή θα πρέπει να ισχύσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η σχεδόν ολοκληρωτική εξάλληψη της γραφειοκρατίας. Το κόστος της γραφειοκρατίας είναι σημαντικό. Σχεδόν τόσο υψηλό όσο και το κόστος των επενδύσεων. Η αηφόρος ανάπτυξη, για να απαντήσω στους διάφορους συναδέλφους που ρώτησαν γι' αυτό, προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις είναι η εφόρος ανάπτυξη να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις ε, που καταναλώνουν και να γίνει πιο εύκολη, πιο ευέλικτη τόσο από άποψη αδειών όσο και από άποψη ε, κάλυψης ε, ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα οι καταναλωτές είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Μια μεγάλη επιχείρηση που έχει σημαντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό της για ενεργειακή ηλεκτρική κατανάλωση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται ακόμη και αν αυτή η ενέργεια παράγεται σε άλλο τόπο από εκεί όπου βρίσκεται η επιχείρηση επειδή υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην έχει επαρκή χώρο για να παράγει ενέργεια στις δικές της εγκαταστάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπάρξει ευελιξία στις ε, τράπεζες. Είναι λογιστικό το θέμα ουσιαστικά. Αν καταφέρουμε να περάσει αυτή η έννοια, να γίνει κατανοητή, θα αναπτυχθεί βιώσιμα μέσα στον χρόνο αυτός ο τομέας. Επαναλαμβάνω, οι επιχειρήσεις που υπάρχουν στις διάφορες περιοχές δεν χρειάζονται επιχορηγήσεις, χρειάζονται βεβαιότητα των κανόνων και κανόνες που να συνάδουν με τις ιδιαιτερότητες των περιοχών του. Τώρα όσον αφορά τα άτομα και την κατάρτισή τους αυτό είναι απαραίτητο. Αυτός ο τομέας πριν από 7 χρόνια δεν υπήρχε ο τομέας των νεοσημών πηγών ενέργειας. Από όσο ξέρω από την Απούλια πριν από 5 χρόνια καμιά εκατοστή άτομα γνώριζαν τον τομέα. Σήμερα 10.000 άτομα εργάζονται σε αυτό τον τομέα. Το μέρος της κατάρτισης και της διαρκούς κατάρτισης ε, πάνω στη δουλειά είναι πολύ σημαντική. Σίγουρα και το θέμα της εξειδίκευσης είναι σημαντικό, αλλά τα άτομα που εργάζονται σε αυτό το τομέα είναι άτομα που δίνουν νόημα στη λέξη ευφυΐα που είναι, που είναι τόσο της μόδας, το smart, ε, της μόδας σε τόσους πολλούς ε, τομείς. Ε, το ευφυΐς. αυτό παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό το τομέα. Αυτός ο τομέας που σύμφωνα με αυτό που έχω να προτείνω, στο τέλος πρέπει να προωθήσει αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν πλούτο στις περιοχές τους. Πλούτο που βασίζεται στην αηφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εσάς. Εκτός μικροφώνου, κύριε Πρόεδρος. Άκουσα διάφορα με τα οποία συμφωνώ απολύτως, η σημασία δηλαδή που έχουν οι επενδύσεις στον τομέα των δικτύων, στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας, όλα αυτά είναι μέσα τα οποία μειώνουν το κόστος της παραγωγής. Άκουσα επίσης και τα πολύ σημαντικά που υπόθηκαν για τον κοινωνικό διάλογο. Υπάρχει μια συγκριτική, ε, γενικά ένα συγκριτικός πίνακα. βλέπουμε ακριβώς και πώς έχει επηρεαστεί τελευταία το κλίμα του κοινωνικού διαλόγου στην Ισπανία. Έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σαν παράδειγμα στην Ford και στους εργαζομένους έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των γραμμών παραγωγής των εργοστασιών της Ford στην Ισπανία. Είναι ένα παράδειγμα θα έλεγα διαλόγου το οποίο βελτιώνει τις σχέσεις ανάμεσα στην επιχείρηση και τους εργαζομένους και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Τώρα για το πόσο τα μέσα και τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν σωστά ή όχι. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι είναι ανεπαρκή. Εμείς δεν έχουμε μια ουσιαστική βιομηχανική πολιτική από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πάρα πολλούς τομείς στην Ισπανία, σε πάρα πολλούς ενώ παραγωγικούς τομείς, βλέπουμε ότι υπάρχει η διαφορετική ε, μεταχείριση ανάμεσα στις απαιτήσει οι οποίες υπάρχουν από τη μία και στις απαιτήσει που εμείς οι ίδιοι ε, περιπτώσει έχουμε απέναντι στις, ε, σχετικά με τις ανάγκες και την χρηματοδότηση την οποία θα μπορούσαμε να είχαμε. Κάτι άλλο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το πόσο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε τομείς δημοσίων ε, επενδύσεων και σε επίπεδο δημοσίων προμηθειών ε, εφόσον πρόκειται να γίνονται επιλογές, με ποια κριτήρια θα γίνονται οι επιλογές των επιχειρήσεων και τι ρόλο θα παίζει ο τοπικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία. Αν θέλουμε πράγματι εμείς να βοηθήσουμε την διατήρηση της παραγωγής στη χώρα και να χρησιμοποιήσουμε φυσικά και μέσα όπως η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, έχει μεγάλη σημασία να να υπάρξει μια συνεκτικότητα απέναντι στις επιχειρήσεις και σε σχέση με τις επιλογές. Γιατί επαναλαμβάνω ότι η πολιτική των δημοσίων προμηθειών είναι εν μέρη μια πολιτική επενδύσεων και είναι σημαντικό κομμάτι της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας μας. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και γι' αυτό θα απαντήσω ίσως στις τέσσερις πιο σημαντικές από τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Πρώτον, σχετικά με το 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ για την έρευνα κτλ. Ε, αυτό ξέρουμε ότι πολιτικά είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τι εναλλακτική λύση υπάρχει. Η εναλλακτική λύση είναι να αφήσουμε τα πράγματα όσοι έχουν, ε, συνεχιζόμενη φτώχεια, αναπτυσσόμενες ανισότητες, απειλή στην επιβίωση του Euro. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το 2% του ΑΕΠ πρέπει να το επιδιώξουμε γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο μεν πολιτικά αλλά έτσι θα μπορέσουμε νομίζω να πετύχουμε κάποιες άλλες πολιτικές αναλλακτικές. Και εδώ νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα για τις ικανότητες και τα προσόντα των εργαζομένων. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει επένδυση στον τομέα αυτό. Να αναφερθώ στο ότι αν πράγματι θέλει κανείς να επενδύσει στον τομέα αυτό, τα, οι συλλογικέ συμβάσεις και οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί μπορεί να υπάρξουν συνολικές αποφάσεις οι οποίες είναι εύκολα εφαρμόσιμες. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε και τις ε, προσωρινές μορφές απασχόλησης, διότι οι προσωρινές μορφές απασχόλησης δεν συνοδεύονται από σωστή κατάρτιση. Τι βλέπουμε όπως τον νότο της Ευρώπης, καταστροφή των συλλογικών συστημάτων διαπραγμάτευσης, και αύξηση των προσωρινών μορφών απασχόλησης. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και να γνωρίζουμε τους κινδύνους. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι, ε, είναι όμοιρος των αγορών. Αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την τράπεζα είναι ότι ανησυχεί για το 3α της βασικά η τράπεζα αυτή και την πρόσβασή της σε φθηνές πιστώσεις στην αγορά. Αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό τότε θα υπάρχουν τα προβλήματα στα οποία εσείς αναφερθήκατε. Γιατί από τα 60 δις που είχαν αποφασιστεί να χρηματοδοτηθούν από, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μόνο τα 15 έχουν ε, αρχίσει να δαπανώνται. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χαμηλώσει το βαθμό μόχλευσής της και έτσι θα δώσει αξιοπιστία στο 3α της. Τώρα για τον κοινωνικό διάλογο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ακριβώς την ε, ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η Ευρώπη μπορεί να ειδωθεί σαν μια προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα. Είναι ένας τρόπος να βλέπει κανείς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι από το 1990 και μετά ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε η εσωτερική αγορά και ε, ε, τότε υπάρχουν και ανάπτυξη ανταγωνισμού ανάμεσα στις οικονομικές πολιτικές και στις ε, εργασιακές ρυθμίσεις και η κρίση οικονομική χρησιμοποιήθηκε ε, σαν άλοθη για την ενίσχυση περαιτέρω του οικονομικού πυλώνα. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν είναι ένας οικονομικός πυλώνας πανίσχυρος ο οποίος στην ουσία σκιάζει και θα υπονομεύει και θα σβήσει τον κοινωνικό πυλώνα. Αν πράγματι θέλει κανείς να, έχει, να υπάρχει κοινωνικός διάλογος και αν πράγματι θέλουμε ο κοινωνικός διάλογος να είναι αποτελεσματικός, κάτι θα πρέπει να γίνει σχετικά με την επανεξισορρόπηση του κοινωνικού με τον οικονομικό πυλώνα. Ευχαριστούμε και για αυτές τις ε, σκέψεις. Ας περάσουμε στο τρίτο πάνελ εντάχει. Ζητώ συγγνώμη από τους ομιλητές, αλλά πάντα συμβαίνει αυτό στο τέλος. Ε, ο χρόνος είναι λίγο πιο περιορισμένος. Έχετε 10 λεπτά. Θα θυσιάσουμε το χρόνο των ερωτήσεων για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε στις 12.30 που είναι το αναποφευκτό όριο. Μιλήσαμε για τους πόρους, Α μιλήσουμε τώρα για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Ας ακούσουμε πρώτα τον Ντάνιελ Κράους που εκπροσωπεί την Κομφιντούστρια τη Ιταλία. Παρακαλώ. Να σας πω ότι το πρόβλημα της ε, ε, μεταπητικής βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη, όχι μόνο για την ε, βιομηχανία, αλλά για την ευημερία όλη τη Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να το παραδεχτούμε ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, τα, με τις δραματικές συνέπειες της κρίσης δεν έχει αποδώσει ακόμα τους καρπούς που θα έπρεπε να έχει ε, αποδώσει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το παραδεχτούμε και να το αναγνωρίσουμε. Τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσει την κρίση ε, εξυπηρετούν όλα από τον ίδιο σκοπό, την ε, διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών. Αλλά δεν έχουν πάρει υπόψη ποιε είναι οι συνέπειε που θα έχουν αυτά τα μέτρα στην οικονομία. Και μέσα σε αυτά τα μέτρα λοιπόν είναι αυτή η άνευ προηγουμένων ύφεση για τη σταθερότητα των δημοσιονομικών φυσικά αποτελεί ένα στόχο πέρα από κάθε αμφιβολία. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως και τις αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις πολιτικές που επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στη λιτότητα. Στην συζήτηση λιτότητα εναντί ανάπτυξης θα πρέπει να βρούμε τα στοιχεία για μια πιο ισόρροπη προσέγγιση που θα συμφελιώσουν την ε, στεναρότητα της οικονομίας με την ανάπτυξη της και θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντα την ε, ανάκαμψη της ε, ανάπτυξης και να γίνουν ανάλογες προσπάθειες δίνοντας μια νέα όθηση στην οικονομία και δίνοντας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τους νέους ιδιαίτερα και νομίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται η ανακοίνωση για την ανάπτυξη και όλες οι προσπάθειες που γίνονται προκειμένου να τοποθετηθούν στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών δράσεων οι πολιτικές αυτές. Αλλά χωρίς καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση δεν θα πετύχουμε πολλά. Γιατί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά για επιτυχή βιομηχανική πολιτική. Και είναι κρίσιμη σημασία για τις ε, επιχειρήσεις και για την οικονομική ανάπτυξη να υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αυτό έχει να κάνει με την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις σχετικές επενδύσεις. Ε, τις τελευταίες μήνες οι, ανά... οι πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί δραματικά. Ενώ τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων συνεχίζουν να είναι διαφορετικού ύψους ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τις χώρες όπου ετούνται τραπεζικό δάνειο επιχειρήσεις. Για να καταλάβετε, τα επιτόκια για βραχυπρόθεσμα δάνεια επιχειρήσεις το Φεβρουάριο του 2013 κειμενόταν στο 5,2 στην Ισπανία και στο 4,4 στην Ιταλία σύγκριση με το μέσο όρο του 3,8 στην Ευρωζώνη. Ως αποτέλεσμα, πολλές επιχειρήσει, ειδικότερα σε περιφερειακέ οικονομίες όπως τι οικονομίε τη Νότια Ευρώπης, αποκλείστηκαν από τραπεζικά κονδύλια, ανεξαρτήτως ποιότητας των επιχειρηματικών τους έργων. Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα από άλλες πηγές όπως επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες ε, μειώθηκαν επίσης σημαντικά κατά την κρίση και μάλλον θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα λόγω του αβέβαιου οικονομικού κλίματος ε, και τους νέους ε, χρηματοοικονομικούς κανονισμούς. Εκτός από τις επιπτώσεις για τα εταιρικά οικονομικά, επηρεάζονται επίσης και τα οικονομικά των εξαγωγών, καθώς και επενδύσεις σε υποδομές που απαιτούν υψηλά κεφάλαια, όπως μεταφορές και τηλεπικοινωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο Υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν πρώτα απ' όλα. Οι μεταρρυθμίσεις των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών θα πρέπει να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης της οικονομικής σταθερότητας και, της, και των οικονομικών αναγκών των εταιριών. Αυτό θα απαιτήσει σωστό υπολογισμό των παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών ώστε να μην δημιουργηθούν νέες αρνητικές επιπτώσεις για τη βιομηχανία. Πιστεύω ότι όλη η συζήτηση για το Βασιλεία 3 δείχνει ότι επιβάλλονται από κάποιους κανόνες μεγαλύτερες κυρώσεις στις μικρότερες βιομηχανίες από τις μεγαλύτερες. Επιπλέον, μια ανάπτυξη συγκεκριμένων εναλλακτικών ε, χρηματοδοτήσεων από τις παραδοσιακές τραπεζικές θα πρέπει να βρεθεί και να υποστηριχθεί. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ελάχιστη ε, πρόσβαση στις κεφαλαίες αγορές. Τα μέτρα δημιουργίας αγοράς θα πρέπει να επικεντρώνονται στη βελτίωση της διαφάνειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση των κινδύνων καθώς και στην αντιμετώπιση του κόστου συναλλαγών δεδομένων των χαμηλότερων ασφαλιστικών δικλείδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η διάδοση των βελτιστών πρακτικών όσον αφορά την καθιέρωση αγορών ομολόγων που να στις οποίες να έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους θα παίξει σημαντικό ρόλο. Τα κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου είναι ένα άλλο σημαντικό χρηματοοικονομικό εργαλείο από μακροοικονομική άποψη. Προς το παρόν οι σχετικές εταιρείες ε, διαδραματίζουν ελάχιστο ρόλο ως πηγή. Οι ασφαλιστικές εταιρείε παίζουν ελάχιστο ρόλο ως ε, πάροχη κεφαλαίων ε, υψηλού κινδύνου. Ενώ στις ΗΠΑ συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο με τα κατάλληλα πλαίσια, φορολογικά κίνητρα για τα κεφάλαια υψηλού κινδύνου και με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές θα μπορέσουν να γίνουν συμμαχοί μας τα νέα χρηματοοικονομικά μέσα που χειρίζονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα διευκολύνουν την παροχή πιστώσεων και τη χρηματοδότηση δεδομένης αυτής της θετικής εμπειρίας πρέπει οπωσδήποτε να ε, βρούμε τα νέα διάδοχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Horizon. Τέλος θα ήθελα να τονίσω συμπεραίνοντας ότι για να είναι επιτυχής μια πολιτική, μια βιομηχανική πολιτική, απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση. Όσον αφορά τη συμφωνία που επιτευχθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Φεβρουάριο, τα σήματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Το επίπεδο δαπανών για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί ιστορική πτώση σε σχέση με τους υπόλοιπους προπολογισμού παρά τις όποιες περικοπές οι αποφάσεις ε, κατανομής των πόρων τουλάχιστον θα έπρεπε να δείχνουν κάποια συνοχή με τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ευθυγραμμίζονται με τον ρόλο που θα διαδραματίσουν επενδύσεις για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κράους για την παρουσίασή σας. ο έχει λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να πάρω το λόγο σήμερα μπροστά σας. Θα συμφωνήσω εν πωλής για αυτά τα οποία, με αυτά τα οποία είπε ο Δόκτωρ Κράους. Ακούω εδώ, ε, εδώ και μια μισή ώρα τις ομιλίες και θα ήθελα λίγο να παίξω το ρόλο του δικηγόρου του διαβόλου. Ε, να πούμε ότι η λύση στα προβλήματα, σε όλα τα προβλήματα δεν είναι η εκβιομηχάνηση. Θυμάμαι πριν πέντε χρόνια όταν πραγματικά όλοι ε, γελιοποιούσαν το γερμανικό μοντέλο και όλοι πίστευαν ότι το μέλλον είναι στις υπηρεσίες. Το θέμα είναι σοβαρό, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Υπάρχουν κάποιες ε, μη παραδοσιακές βιομηχανίες εκτός του τομέα των υπηρεσιών, που καλούνται να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της ανάκαμψης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν αυτούς τους τομείς της οικονομίας, γιατί είναι κρίσιμοι τομείς για την οικονομία. Και ο τομέας των υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικός και δεν θα πρέπει βέβαια να τον αγνοήσουμε. Λοιπόν τώρα, έρχομαι στο θέμα που μας απασχολεί σήμερα για την αποβιομηχάνηση στο νότο της Ευρώπης και τις νέες δυνατότητες εκβιομηχάνησης. Εγώ ξεκινώ θα έλεγα με τα βασικά μηνύματα που θα ήθελα να μεταφέρω. Το νότος και το κέντρο της Ευρώπης έχουν σημειώσει μια από εκβιομηχάνηση οδηγό ε, προς την κρίση χρονικά. Σαν παράδειγμα είναι η Γαλλία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κάποια πρόοδος βέβαια σε σχέση με την αύξηση των εξαγωγών. Αυτό δείχνει ότι έχουμε αρχίσει να βλέπουμε μια μετακίνηση στην διάρθρωση των προτύπων παραγωγής στις διάφορες χώρες. Τρίτον, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θα έλεγα διαρθρωτικά εμπόδια στην ανάπτυξη της βιομηχανίας Κυρίως θα πρέπει να σταθούμε στα θέματα της χρηματοδότησης βέβαια και να πούμε ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα τεράστιο θέμα και το έχετε υπογραμμίσει αυτό όπως και ο κύριος Κράους. Αλλά θα σας δείξω κάποια slides που να αποδεικνύουν την μεγάλη σημασία αυτής της ελλειπούς χρηματοδότησης απαραίτητης για την αποκατάσταση των προβλημάτων στην Νότια Ευρώπη. Βλέπετε, έχετε ήδη δει τον πίνακα αυτό, βλέπετε ακριβώς ε, τη μείωση της μεταποιητικής δραστηριότητας στις διάφορες χώρες, ε, Ελλάδα, Ιταλία, ε, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία. Βλέπετε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, αλλά έχει υπάρξει μια ουσιαστική μείωση της εκβιομηχάνησης. Βλέπετε όμως ότι η μείωση αυτή τα τελευταία χρόνια μάλλον έχει σταματήσει. Δεύτερον, βλέπετε επίσης το κέντρο εδώ που είναι η Γαλλία, όπου υπήρξε μια πιο σημαντική μείωση στον τομέα της μεταποίησης. Εδώ έχουμε έναν ενδιαφέροντα πίνακα, ο οποίος ασχολείται με, τα, με τις συνιστώσεις που εξηγούν τις αλλαγές στο ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, περίοδος 2007-2012. Λέγεται γενικά ότι η μείωση προέρχεται από τη μείωση της ζήτησης. Ε, παίζει ρόλο βέβαια στις αλλαγές αυτές ε, η μείωση της ζήτησης, αλλά και οι εξαγωγές παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να υπάρξει μια κάποια ρύθμιση των εξωτερικού τύπου έλλειψης ισορροπιών. Νομίζω ότι πολλές φορές οι εξαγωγές είναι ε, κατευθυντήρια γραμμή και δύναμη για την αποκατάσταση της ισορροπίας σε χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιταλία. Ε, οι τρέχουσες συναλλαγές στην Ελλάδα επηρεάζονται από την μείωση κυρίως, τη συντριπτική μείωση των εισαγωγών και η εξαγωγική δραστηριότητα δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την ισορροπία των τρεχουσών συναλλαγών. Τώρα για, τις, για τα διαφθρωτικά εμπόδια, τρία είναι τα βασικά σημεία. Πρώτον, στα θέματα της έρευνας που έχει κάνει και το Ινστιτούτο Μπρούγκελ σχετικά με το τι οδηγεί την ανταγωνιστικότητα και τι οδηγεί τις επιδόσεις στον τομέα των εξαγωγών. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο ανέπτυξε ο Ταβιάνο και ο Αντιμόντι. Ένας από τους παράγοντες τον οποίο εντόπισαν είναι ότι είναι σημαντικό για τη βιομηχανία να μπορεί να εξάγει ανάλογα με το μέγεθος. Απαιτείται μεγάλο μέγεθος για να μπορεί να εξάγει κανείς, απαιτείται να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να γίνει ανταγωνιστικός. Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί πολλές χώρες στο νότο της Ευρώπης οι επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες έχουν ε, μικρό μέγεθος γενικά. Τίθεται λοιπόν ένα θέμα και εδώ υπάρχουν και προβλήματα νομικά που επιβαρύνουν την κατάσταση. Κάποιοι ε, βλέπω ότι δεν μπορεί να διαβαστεί εύκολα αυτός ο πίνακας, αλλά η τρίτη στήλη βλέπετε ότι είναι σχετικά κόκκινη σε σχέση με τις υπόλοιπες στήλες σε σχέση με ορισμένους δείκτες όπως αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, επιχειρηματικότητα, ρύθμιση των αγορών κτλ. Βλέπουμε ότι οι παραδοσιακοί δείκτες δείχνουν ότι ο νότος της Ευρώπης πηγαίνει χειρότερα από ότι ο βορράς της Ευρώπης. Κάτι το οποίο δείχνει και εξηγεί τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Τώρα σχετικά με το χρηματοδοτικό κομμάτι. Όλοι γνωρίζουμε τις δραματικές ε, διαφορές σε σχέση με τα ομόλογα τα κρατικά και τα δικαιώματα δανεισμού. Αλλά έχει υπάρξει όμως από το προηγούμενο καλοκαίρι μια μείωση αυτού του κενού, αυτής της διαφοράς ανάμεσα στα επιτόκια δανεισμού. Παρόλα αυτά ποικίλουν στο εσωτερικό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγκάζονται οι κυβερνήσεις να πληρώνουν πάρα πολύ ψηλά επιτόκια. Ε, στις αγορές των κρατικών ομολόγων είναι το κατώτερο επίπεδο σε σχέση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης της βιομηχανίας. Δηλαδή, αν το εξωτερικό χρέος, το δημόσιο χρέος είναι σε κακή κατάσταση, τότε πολύ συχνά επηρεάζεται άμεσα, άσχημα, η βιομηχανική δραστηριότητα. Υπάρχει επίσης και το θέμα του ε, τραπεζικού συστήματος το οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα. Εδώ να σας δείξω ε, για τα μη αποδοτικά δάνεια. Βλέπετε εδώ τις χώρες που μας ενδιαφέρουν. Βλέπετε ότι έχουν αυξηθεί τα δάνεια αυτά τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει σαφώς την δυνατότητα των τραπεζών να μπορέσουν να δανείσουν με βιώσιμο και χρήσιμο τρόπο. Τα πιστοτικά προβλήματα λοιπόν είναι κεντρικά προβλήματα στην προσπάθεια της αποκατάστασης των οικονομικών συνθήκων για την ανάπτυξη της Νότιας Ευρώπης. Τώρα, πάντα στα θέματα της χρηματοδότησης είναι, είναι τα επιτόκια, τα ύψη των επιτοκίων. Εδώ βλέπετε ότι το χαμηλότερο, το κόκκινο, είναι η Γερμανία. Αυτό που δείχνει αυτή η διαφάνεια είναι ότι οι χαμηλές πιστώσεις μπορεί να είναι πολύ πιο ευθυνές στην Γερμανία παρότι στο Νότο. Και αυτό είναι ένα συγκριτικό μειονέκτημα ε, για τον Νότο. Τέλος, δεν είναι μόνο τα επιτόκια, αλλά και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Εδώ βλέπετε το ποσοστό των αιτήσεων και των ποσών που έχουν εγκριθεί ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή ζητούν πίστοση οι μικρομεσαίες ε, και τους δίδεται η πίστοση αυτή. Ποιο είναι το ποσοστό των θετικών λοιπόν αποκρίσεων των τραπεζών. Βλέπετε ότι η Γερμανία είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Όλες οι μικρομεσαίες παίρνουν δάνεια αν πάνε σε μια τράπεζα και τα ζητήσουν ενώ οι πέντε χώρες του Νότου κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Στην Ελλάδα μόνο το 25% εγκρίνεται των ετοιμάτων. Αν ε, θέλετε να κάνετε μια επιχείρηση στην Ελλάδα και πηγαίνετε στην τράπεζα, τότε έχετε 25% πιθανότητα να πάρετε το δάνειο. Πάρα πολύ χαμηλό. Το θέμα είναι και ποιοτικό και ποσοτικό βέβαια. Τώρα υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υποσυζήτηση και πάνω στα οποία γίνονται κάποιες μελέτες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σαν παράδειγμα, έχει προβλέψει ένα, πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί 15 δις. Γίνονται κάποιες προσπάθειες επίσης και από το Γενικό Κρατικό Λογιστήριο και το αντίστοιχο Γερμανικό και τη Γερμανική Δημόσια Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε να τονωθεί η, ε, η ε, δραστηριότητα και η δυνατότητα δανειοδότησης στην ε, Νότια Ευρώπη. Έχει γίνει μια τέτοια προσπάθεια και για την Πορτογαλία. Δείτε όλους αυτούς τους αριθμούς θα καταλάβετε σαφώς ότι μιλάμε για μικρά ποσά. Και στην καλύτερη περίπτωση είναι μια σταγόνα αν θέλετε στον ωκεανό και δεν βοηθούν πάρα πολύ. Δεν βοηθούν αρκετά. Το μεγάλο πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται υποσυζήτηση στην παρούσα φάση είναι το τι πραγματικά θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι ώστε οι τράπεζες που δανείζουν στις μικρομεσαίες να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν ευθυνότερη ρευστότητα ή μικρότερη επιβάρυνση εν πάση περιπτώσει. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι σε επίπεδο τεχνικό η προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, πάντως παραμένει ένα από τα σημαντικά κεντρικά θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να αποκατασταθεί ο μηχανισμός, ε, ε, να αντικατασταθεί ο μηχανισμός ρυθμίσεων των προβλημάτων και των αποκλήσεων μέσω των νομισματικών πολιτικών. Ε, πάντως δεν υπάρχει εδώ πολλά, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία επίσης στους ισολογισμούς των πιστοτικών ιδρυμάτων και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Δίνω τον λόγο στον κύριο Μπουτικόφερ για να κάνει την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστούμε και τους δύο μελητές ε, για τις παρουσιάσεις τους. Έχω δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτα προς τον κύριο Βόλφ. Συμφωνείτε με τη θέση του συναδέλφου του κύριου Κράους όσον αφορά αυτό που ονομάζει ανάγκη επαναβαθμονόμηση των μεταρρυθμίσεων στον οικονομικό τομέα, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει πιο ευρία χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, το οποίο εγώ μεταφράζω, όπω έχουμε ξανασυζητήσει παλιότερα με την κομφιντούστρια, το μεταφράζω σε φρενάρετε το Basel 3 για να διασφαλίσετε περισσότερο δανεισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Δεύτερον, κύριε Κράους, αναφέρατε τις αγορές ομολόγων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα παράδειγμα στη Στουτγάρδη που λειτουργεί πολύ καλά. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια ώστε να προωθήσει τέτοια παραδείγματα και τέτοιες πολιτικές. Και προς τους δυο σας υποστηρίζετε την πρόταση που ακούστηκε νωρίτερα ότι θα έπρεπε να έχουμε μια ενιαία αγορά κεφαλαίων ε, ε, υψηλού κινδύνου στην Ευρώπη, τα venture capitals και ποια θα ήταν τα πρακτικά βήματα που πρέπει να κάνουμε για αυτό το σκοπό. Και τέταρτον, η διασφάλιση δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα που ανέφερα στην αρχή και με τα διευθυντικά ομόλογα. Για ποιο είδου μικρομεσαίε επιχειρήσει θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί, Είναι πρακτική πρόταση, βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λύση. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, πριν ξαναδώσω το λόγο στους δύο εισηγητές του Παναλαυτού, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Γενικής φύσης μάλλον, αλλά που είναι μια ερώτηση που απασχολεί όλους μας δεδομένης της δυσκολίας πρόσβασης σε πιστώσεις ή της περιορισμένης πρόσβασης της πιστώσης ή της υπερβολικά ακριβής πρόσβαση σε πιστώσεις, αιτίες που συχνά οδηγούν σε διακοπή μιας παραγωγικής δραστηριότητας. Τι θα μπορούσαν να κάνουν ακόμη πέραν των όσων είπατε η Κεντρική Τράπεζα και η Επενδυτική Τράπεζα. Δεν μιλάω για ένα μαγικό ραβδάκι, απλά ποιες θα ήταν οι δυνατότητες ε, δεδομένων των περιορισμών που έχουμε σήμερα, τι θα προτείνατε να γίνει. Και μετά πώς εξηγείται σε αυτό το μυστήριο στην Ευρώπη όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, παρέχει σε ορισμένες χώρες ε, δάνεια με πολύ χαμηλά επιτόκια σχεδόν ανύπαρκτα και ότι όταν αυτό το, αυτή η πίστοση φτάνει υπό την μορφή δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα επιτόκια είναι πολύ ψηλότερα και όλοι διαμαρτύρονται ο πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων, ο πρόεδρος Κομισιόν, η οικονομική υπεύθυνη των κρατών μελών, αλλά κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Όταν εμένα ένας ψηφοφόρος με ρωτάει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Δεν θα μπορούσε να δοθεί ένα κομμάτι αυτών των πιστώσεων πιο φθηνά πώς θα μπορούσε, από ποιον εξαρτάται το να δοθούν αυτές οι πιστώσεις ε, με επιτόκια χαμηλότερα. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο, ε, πάρτε το λόγο με το σειρά που θέλετε εσείς. Try to, to Να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που ακούσαμε. Πώς δημιουργούμε μία ε, έγκυρη αγορά μετοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι Μόνο με τους κατάλληλους και αυστηρούς κανόνες μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη δράση σε κάθε κράτος μέλος. Ιδάλλως θα έχουμε μεγάλες διαφορές και μια κατακριματισμένη αγορά. Συγκεκριμένες δράσεις λοιπόν. Και θεωρώ ότι θα πρέπει και οι ευρωπαϊκές τράπεζες να οραματιστούν, αν θέλετε, την ε, δημιουργία αυτής της αγοράς. Κατά δεύτερον, δεύτερο ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει μία ενιαία αγορά για τα επιχειρηματικά κεφάλαια και θα έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή. Ναι, φυσικά. Πότε λειτουργεί καλά η αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων όταν η οικονομία είναι μεγάλη, όπως της είπα. Είναι η έκταση, η διάσταση αυτή που παίζει σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο ο αριθμός των επιχειρήσεων, αλλά και ο όγκο σε ό,τι αφορά τη διάδραση μεταξύ των τομέων. Άρα η Ευρώπη δεν μπορεί να το αφήσει αυτό στην ευχαίρεια του κάθε κράτους μέλους. Η Ευρώπη θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ενθαρρύνει τις ε, αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Προκειμένου να ενθαρρύνει και τους επενδυτές. Ακόμα και οι χώρες όπως ε, η Ινδία, για παράδειγμα, σήμερα δίνουν κίνητρα σε επενδυτές στην αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων. Γιατί λοιπόν η Ευρώπη να μην κάνει το ίδιο. Να απαντήσω στο ότι συμφωνώ. Θεωρώ ότι για να ασφαλιστεί η αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων για, τα, για τις πιστώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μια λύση γιατί θα πρέπει να βρεθεί ένα πλαίσιο για την πρόθεση της λύσης αυτής. Και νομίζω ότι και εδώ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να απαντήσω όμως και το τελευταίο ερώτημα που έθεσε η κυρία Τόγια. Πολύ σχετικό ερώτημα θεωρώ ότι σήμερα, ιδιαίτερα στην ε, Νότια Ευρώπη, από ό,τι είδαμε από την παρέμβαση του κυρίου Βόλφ, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την ε, τιμή των πιστώσεων, αλλά και την διαθεσιμότητα των πιστώσεων, γιατί στη Γερμανία 90% των επιχειρήσεων που έχουν ε, κάνει αίτηση για πίστοση λαμβάνουν την πίστοση αυτή, ενώ στην ε, Ισπανία το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 60% στην Ελλάδα μέχρι και 30%. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα διαθεσιμότητα. Ασφαλώς οι τράπεζες ακολουθούν τις παλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την θεσιμότητα των πιστώσεων, αλλά οι τράπεζε νομίζω ότι είναι πολύ διστακτικέ στην χορήγηση δανείων, γιατί πολλοί από του ετούντε για δάνεια έχουν σημειώσει αποτυχίες, αν θέλετε, ή δραστηριοποιούνται σε τομείς που έχουν πληχθεί ιδιαίτερως από την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουμε τις τράπεζες, ε, εξηγώντα τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές σε ό,τι αφορά εταιρικά δάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική από πλευράς της Ένωσης σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις πηγές εναλλακτικής ε, ενέργειας. Κατά το παρελθόν, πολλές ε, εταιρείε που παρήγαγαν ηλιακά πάνελ και έλαβαν πιστώσεις από τις τράπεζες για την παραγωγή των πάνελ αυτό, πλέον ε, τους τα φέρουν τα δάνεια, τους τα ζητούν πίσω. Αυτό αποτελεί απόρρια ε, της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κινέζικου dumping, dumping και οι επιδοτήσεις δεν είναι παρόμοιες με αυτές των Αμερικανών. Άρα αφενός λέμε ότι θα πρέπει να δώσουμε να τονώσουμε την παραγωγή, γιατί η παραγωγή είναι πάρα πολύ σημαντική και την υποστηρίζουμε, αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την χρηματοδότηση αυτών των νέων κατασκευών. Νομίζω ότι το θέμα των πιστώσεων σχετίζεται ασφαλώς με τις άλλες πολιτικέ. Και εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να δραματίσει το ρόλο του έναντι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τι πολύ σημαντικέ ερωτήσει που θέσατε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω για το ζήτημα του Βασιλεία 3. Το ζήτημα που θέτεται είναι εξαιρετικά περίπλοκο και μας απασχολεί ιδιαίτερος. Θα προτιμούσα να απαντήσω πιο γενικά θα σας μιλήσω γενικά, διότι οι ιδιαιτερότητες του Βασιλεία 3 είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Από γενική άψη λοιπόν, το τραπεζικό μας σύστημα αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες επίσης λόγω του γεγονότος ότι υπήρχαν ανεπαρκή κεφάλαια στο τραπεζικό σύστημα και αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Συνεπώς, ο στόχος αύξησης των κεφαλαιακών επιπέδων εντός του τραπεζικού συστήματος είναι πολύ σημαντικός στόχος και δεν πρέπει να τον παραβλέπουμε διότι χωρίς ε, ένα πιο σταθερό και ένα πιο οικονομικά υγιές ε, τραπεζικό σύστημα υπάρχει κίνδυνος να την πληρώσει ξανά ο φορολογούμενος όπως έχει συμβεί μέχρι σήμερα και ακόμη περισσότερο πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε την οικονομική κρίση όπως αυτή που είδαμε πρόσφατα. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο στο τραπεζικό σύστημα. Μπορεί να συζητήσει βέβαια κανεί το πόσο χρειάζεται, ποια στιγμή πρέπει αυτό να ε, δοθεί και πώ. Αλλά ο στόχο αυτό είναι απολύτω κρίσιμη σημασία. Εγώ λοιπόν ε, δεν θα υποστήριζα το να αποδυναμώσουμε το Βασιλεία 3 στην παρούσα φάση. Ας το καθυστερήσουμε ίσως λίγο, αλλά λόγω των χρηματοδοτικών συνθήκων αυτή τη στιγμή στο τραπεζικό σύστημα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκοπός πρέπει να είναι να ε, εισάγουμε περισσότερο κεφάλαιο στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό ίσως σχετίζεται ίσως και με την τελευταία ερώτηση, τη δική σας ερώτηση κυρία Πρόεδρε για το τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Θα ήθελα να εκφράσω την επιφύλαξή μου όσον αφορά τη δυνατότητα τα δημόσια τραπεζικά ιδρύματα να αντικαταστήσουν τα ιδιωτικά. Αυτό είναι αδύνατο. Το τραπεζικό σύστημα είναι τεράστιο. Γνωρίζει τους πελάτες, γνωρίζει ποιοι είναι σωστοί και όχι πιστωτές. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την ε, ενισχυμένη ίσως κεντρική τράπεζα της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να κάνουμε είναι να είναι βιώσιμο τραπεζικό μα σύστημα και να μπορεί να παράσχει πιστώσεις στις τράπεζες. Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και ένα σημαντικό είναι οι διαφορετικές συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά σχετίζονται με το όλη συζήτηση περί Τραπεζικής Ένωσης. Κατά την άποψή μου λοιπόν το σημαντικότερο που πρέπει να επιτευχθεί εδώ είναι μια πλήρης, ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση που θα επιτρέπει στις τράπεζες, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται, να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε ίδια κεφάλαια και συνεπώς να μπορούν να παράσχουν πιστώσεις σε επιχειρήσεις. Τέλος, αλλά δύο σημεία όσον αφορά την ενία αγορά κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Συμφωνώ, έχουμε παρατηρήσει μια τεράστια μεταβολή στο τραπεζικό μα σύστημα από τις τράπεζες προς ε, χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβήτες ε, άλλου τύπου, αλλά πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή είναι καλή και θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτή την παρέμβαση που να βασίζεται σε κεφάλαια και χρειαζόμαστε φυσικά μια κεφαλιακή αγορά υψηλού κινδύνου καθώς και τα ε, ομόλογα για τα οποία συζητήσαμε. Τέλος όσον αφορά την ε, διασφάλιση, το ανέφερε νομίζω ο κ. Μπιούτικοφ, η διασφάλιση των δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει γρήγορα και είναι βιώσιμη λύση. Εγώ πιστεύω ναι, μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί Το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια δημοσιονομική διάσταση. Όσο περισσότερο κάνει μια τράπεζα κάτι τέτοιο, τόσο χαμηλώνοντα για παράδειγμα τα πρότυπα εγγύσεων, τόσο περισσότερου κινδύνου αναλαμβάνει κανεί όσον αφορά τον ισολογισμό τη ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα, αν τα πράγματα ήταν ιδανικά, θα μπορούσε κανεί να το κάνει αυτό και να έχει ένα ταμείο από πίσω, όπω γίνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε, διότι Εκεί το US Fed αναλαμβάνει όλες τις απώλειες, αλλά εδώ δεν το έχουμε αυτό, συνεπώς τα πράγματα γίνονται λίγα πιο περίπλοκα. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο... ε, Κεντρική Τράπεζα είναι πιο επιφυλακτική να προχωρήσει σε τέτοια ζητήματα. Αν θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει, όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστεί το δημοσιονομικό ζήτημα είτε με μια συμφωνία του Eurogroup να καλύπτονται οι χρηματικές ε, ζημίες ή κάτι τέλος πάντων. Εάν το θέλουμε, εάν είναι επιθυμητό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό ακόμα κύριε Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά μου ζητήσατε ένα λεπτό θα του το παράσχουμε και ζητώ από τους διερμηνείς ένα λεπτό παράταση. Πιστεύω ότι οι τράπεζες και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου είναι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Εμείς στις Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούμε ότι πρέπει να κινητοποιούμε ιδιώτες με πολλά χρήματα να ρίψουν κινδυνεύσουν επενδύοντας σε νέους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει η Ευρώπη. Δείτε το παράδειγμα του Ισραήλ. δείτε αυτή την προσέγγιση του Ισραήλ που είχε μεγάλη επιτυχία για τους νέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων και ειδικότερα εκ μέρους του κυρίου Σύγητη του κυρίου Μποτικόφερ όλους τους ομιλητές σήμερα το πρωί. Δεν χρειάζεται να καταλήξουμε συμπεράσματα διότι όσα είπατε θα οδηγήσουν σε σκέψεις και προβληματισμό και σε μελέτη κατά τις εργασίες μας. Αυτό είναι πιστεύω το καλύτερο συμπέρασμα Ευχαριστούμε για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και ευχαριστούμε και τους συναδέλφους που παρέστησαν εδώ.